Vamos Λοιπόν, ας ξαναρχίσουμε τις εργασίες μας. Θα ξεκινήσουμε από το σημείο 16. Αναφορά 1274 του Λίους Πένιο Κάγιος Μποένο, Ισπανικής καταγωγή του νόμου της Επιτροπής Ερμίλ, σχετικά με τις διακρίσεις που φύστανται οι επιβάτες με αναπηρία από τι αεροπορικές εταιρείες και τον κανονισμό 1107-2006. Λοιπόν, έχουμε και επίση και την 1496-2013 τη Μαρία Ζαμπάρα Απόγεια σχετικά τα δικαιώματα των τόμων με αναπηρή. Θα δώσουμε το λόγο στον εκπρόσωπο ε, των αναφερόντων λοιπόν. Κύριε και κυρίες βουλευτές, ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, κυρία Πρόεδρε, που με επιτρέπετε να πάρω το λόγο. Η ΣΕΡΜΗ εκπροσωπεί τα άτομα με αναπηρία στην ε, Ισπανία. Εκπροσωπεί κυρίως την Εθνική Επικράτεια, είναι πλατφόρμα συνάντησης που προασπίζεται τα συμφέροντα των ανθρώπων με αναπηρία. Το θέμα του σημερινού αφορά τον κανονισμό μέσω του οποίου τίθεται ένα πλαίσιο για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία στις αερομεταφορές, τον κανονισμό ε, του 2006 θα και τον κανονισμό 1107-2006. Θα ήθελα να αναφερθώ και σε κάποιες αρνητικές πτυχές που ε, πλήττουν τα δικαιώματα των ανθρώπων ανεπηρίες για τις αερομεταφορές. Έχουν δυνατότητα οι αεροπορικές εταιρείες να εμποδίσουν έναν ανάπηρο να μπει σε αεροσκάφος ε, προφασιζόμενε ότι είναι θέμα ασφαλείας. Πολύ συχνά τα άτομα με αναπηρία δεν γνωρίζουν τι θα συμβεί ε, με αυτούς, ε, διότι ε, υπάρχουν αεροπορικέ εταιρείε που μπορούν να τους απαγορεύσουν να επιβιβαστούν στο αεροσκάφο. Και μπορεί οι αεροπορικέ εταιρείε να είναι υπερβολικά απαιτητικέ, να θέλουν συνοδό του ανθρώπου με αναπηρία, αλλά ειδή εξόδου. Ε, μπορεί να αποφασίσει η αεροπορική εταιρεία για λόγους ασφαλείας ότι τα άτομα με αναπηρία πρέπει να συνοδεύεται από κάποιον αλλά εις το κόστος είναι εις βάρος του ανθρώπου με αναπηρία πρέπει να πληρώσει για το σύνοδο. Ε, θα πρέπει να ενημερώνουν τουλάχιστον 48 ώρες πριν την πτήση. Τα άτομα με αναπηρία λοιπόν ενοχλούνται, ε, τους εμποδίζεται η κινητικότητά τους και βλέποντας τη Διεθνή Σύμβαση που υπάρχει όσον αφορά τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία που επικυρώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπουμε ότι η σχετική οδηγία εμπεριέχει στοιχεία τα οποία εμποδίζουν τα άτομα με αναπηρία να μπορέσουν να μετακινηθούν και παραβιάζονται κάποια δικαιώματά τους που συμπεριλαμβάνονται στην ελόγω σύμβαση. Το άρθρο 19 της σύμβασης το δικαίωμα για καθολική πρόσβαση που είναι γενική αρχή που επιτρέπει την ε, εφαρμογή των δικαιωμάτων της συμβάσεως. Έχουμε λάβει ε, κάποιες καταγγελίες εδώ μεταξύ άλλων της κυρίας Θαμπαλά Πρόκειται περί ανθρώπου που κινείται με αναπηρικό καροτσάκι και δεν μπόρεσε να επιβιβαστεί εάν δεν συνοδευόταν από κάποιο άτομο ε, που δεν ήταν ανάπηρο. Θεωρούμε ότι αυτή η κατάσταση παραβιάζει τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία, ε, τα δικαιώματα που έχουν ως πολίτες. Και αυτού του είδους τα προβλήματα θα πρέπει να ρυθμίζονται τροποποιώντας τον κανονισμό του 2006 και να υπάρχει πλήρης εγγύηση των δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρία, εμποδίζοντας τις αεροπορικές εταιρείες να απαγορεύσουν την επιβίβαση αυτών, ε, προβάλλοντας ισχυρισμούς ε, περί ασφαλείας. Το αμερικανικό δίκαιο σέβεται περισσότερο ε, τα δικαιώματά τους. Η Αμερικανική νομοθεσία προσθέτει διευκρινήσεις πολύ πιο ευνοϊκές για τα άτομα με αναπηρία ο ευρωπαϊκός εναέριος χώρος και ο, ο αμερικανικός εναέριος χώρος θα πρέπει να αντιβρούν με παρόμοιο ε, τρόπο. Οι υπηρεσίες του check-in online θα πρέπει να υπάρχει, θα πρέπει το προσωπικό επίσης να είναι κατάλληλα καταρτισμένο και ενήμερο. Θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αεροπορικών εταιριών και εκείνων που χειρίζονται τα αεροδρόμια. Η επιβίβαση και αποβίβαση των αναπηρικών πολυθρών θα πρέπει να γίνεται σωστά να μην δημιουργούνται ζημιά και εκεί που προξενεί κάποια ζημιά θα πρέπει να πληρώνει. Το να αρνούνται οι αεροπορικές εταιρείε να επιβιβαστεί κάποιος με αναπηρία και να τον υποχρεώνουν να συνοδεύεται από κάποιον αρτιμελή ε, δεν είναι σωστό. Βρίσκεται ο άνθρωπος με αναπηρία σε μια κατάσταση σαν να είναι υπό την κυδαιμονία κάποιου και παραβιάζεται η σύμβαση του 2006 με αυτόν τον τρόπο. Ο κανονισμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη αυτού του είδους της ε, καταστάσεις και να εξαλειφθεί κάθε διάκριση εις βάρος των ανθρώπων με αναπηρία. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Θα δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ο αναφέρον απευθύνει δύο επικρίσεις σε σχέση με τον κανονισμό. Πρώτον, η υποχρέωση, ή, ε, για να είμαι ακριβέστερος, αναγκαιότητα πρώτερης ειδοποίησης, 7-1 άρθρο του κανονισμού, ε, δεύτερον, η δυνατότητα ε, απόρριψης ε, της επιβίβασης όταν υπάρχει ένα πρόβλημα με το safety, άρθρο 4 του κανονισμού, με την ασφάλεια. για την πρώτερη ειδοποίηση, πρώτερη κοινοποίηση θα πρέπει να γίνεται 48 ώρες νωρίτερα και αυτό ε, και για, ισχύει και για την επιστροφή όταν είναι δηλαδή ε, όταν δεν αποτελείται από ένα μόνο σκέλος ε, το, το, το ταξίδι. Η αεροπορική εταιρεία θα πρέπει στο μέτρο του δυνατού να μεριμνήσει όταν κάποιος με περιορισμένη ε, κινητικότητα υποβάλει αυτό το αίτημα, θα πρέπει να φροντίσει να μερμηνήσει η εταιρεία ούτω ώστε να παρασχεθεί η απαιτούμενη βοήθεια. Βεβαίως υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες ανάλογα με το άτομο. Και με μία ε, πρώτερη κοινοποίηση μπορούμε να εστιαστούμε στις ανάγκες ε, του ατόμου ε, και να μην παρασχεθεί μια γενική βοήθεια, αλλά να ε, παρασχεθεί μια βοήθεια που πραγματικά θα ε, καλύψει τις ειδικέ ανάγκες του συγκεκριμένου ατόμου. Δεύτερον, το δικαίωμα απόρριψη τη επιβίβαση όταν υπάρχει ένα πρόβλημα με την ασφάλεια. Αυτή είναι η δεύτερη επίκριση του ε, αναφέροντος. Άρθρο 7. Όταν υπάρχει πρόβλημα με το άτομο που συνοδεύει, παραδείγματο χάρη, ε, το ΑΜΕΑ. Είναι σαφέστατε οι ρυθμίσεις μέσα στον κανονισμό. Η άρνηση ε, ε, προκύπτει από εθνική και οι ευρωπαϊκές νομοθεσίες σε σχέση με τις διατάξεις ασφάλειας και σχετίζονται με το πιστοποιητικό του αερομεταφορέα και πιο συγκεκριμένα με ε, το μέγεθος ε, της πόρτας της θύρας επιβίβασης ε, και της διαστάσεις του αεροσκάφους. Υποχρεούται ο αερομεταφορέας για το εν λόγω άτομο να προσφέρει μία αποδεκτή εναλλακτική λύση. Αν δεν είναι σε θέση να το κάνει αυτό, θα πρέπει να αποζημιώσει ε, το εισιτήριο, το κόστος του εισιτηρίου ή να ε, βρει μία νέα λύση για ένα νέο δρομολόγιο. Στη συνέχεια πρέπει να γίνει αυτό σε προσβάσιμο μορφότυπο και να δημοσιευτούν οι πληροφορίες και να προσαρμόζονται στις ανάγκες των λόγω ατόμου. Εάν υπάρχει άρνηση θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη και άμεση η απάντηση του αερομεταφορέα. Η αιτιολόγηση θα πρέπει, αν το ζητήσει ε, τον λόγο άτομο, να είναι γραπτή και σε περίοδο πέντε ημερών. Ε, υπό τις ίδιες με που θα ίσχυαν αν ε, υπάρχει ο κανόνας υποχρέωσης συνοδού. Ε, στο μέτρο βεβαίως που ε, ισχύουν αντίστοιχοι κανόνες στη ΕΠΑ. Έχουμε τις κατευθυντήριες γραμμές στις 11 Ιουνίου του 2012, όπου διευκρίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποιες είναι οι υποχρεώσεις στο αερομεταφορέα και μεταξύ των οποίων υπάρχει υποχρέωση άμεση ειδοποίηση ε, του εν λόγω ατόμου κατά την κράτηση ή κατά την πρώτερη κοινοποίηση. Όταν υπάρχει υποχρέωση Συνοδού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ότι ότι θα πρέπει να αιτιολογηθεί αυτό. Αν για λόγους ασφαλείας δηλαδή απαιτείται συνοδός. Εάν όμως δεν προβλέπεται στον κανονισμό θα, θα πρέπει να υπάρξει κάλυψη ε, του ατόμου δωρεάν, χωρίς επιπρόσθετο κόστος. Στη συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει και τις καλές βέλτισες πρακτικές του αερομεταφορέ για όλους τους υπόλοιπους επιβάτες. Nous sommes devant un règlement qui fonctionne bien. Et Επίσης, η πλειοψηφία των ατόμων και οι ενώσεις που αντιπροσωπεύουν τα άτομα με ε, μειωμένη κινητικότητα ικανοποιούνται από τον κανονισμό και οι διατάξεις ε, για την ασφάλεια υπερτερούν κυρίως σε περιπτώσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια ε, του συνόλου των επιβατών ή του πληρώματος δεν προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρηση των λόγων κανονισμό εκ τούτου. Αντίθετα, θεωρεί ότι πάντοτε θα πρέπει για, κατά την εφαρμογή, τη σωστή εφαρμογή του κανονισμού να καταδεικνύουν καλή θέληση οι εθνικές αρχές ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο μέτρο του δυνατού, όπως έκανε και στο παρελθόν, προβαίνει σε διευκρινήσεις των εν Gracias. Eh, tiene la palabra Ευχαριστούμε η Σολεδάδο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, την ε, Σέρμη που είναι παρούσα και παρουσιάζεται ένα θέμα που θεωρώ σημαντικότατο. Πράγματι, Υπάρχει αυτή η πραγματικότητα. Μα λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι επαρκή και γίνεται σεβαστό ο κανονισμό. Αρκεί όμω πιστεύω να ανοίξει κανεί τι εφημερίδε και τα άρθρα για τι αεροπορικέ εταιρείε και κυρίω τι εταιρείε low cost και θα δει ότι όλα τα επιχειρήματα του ΣΕΡΜΗ ισχύουν. θα πρέπει να πληρώνει ε, το κόστος ο συνοδός και πολύ συχνά ε, αρνούνται την επιβίβαση επικαλούμενοι θέματα ασφαλείας. Τα άτομα με αναπηρίες δεν είναι ασθενείς, ίσως χρειάζονται κάποια βοήθεια σε ιδιαίτερες περιστάσεις, αλλά ζουν λίγο πολύ κανονική ζωή και δεν είναι ασθενείς. Οι αεροπορικές εταιρείες δεν πρέπει να επικαλείται θέματα ασφαλείας. Δεν καταλαβαίνω αυτή την ανάγκη επίκλησης ε, ασφαλείας. Και αυτά είναι εμπόδια να πρέπει να προειδοποιεί κανείς πριν 48 ε, ώρες. Και αυτό δεν αφορά την ειδική βοήθεια, η πραγματική βοήθεια. Δεν είναι ασθενείς αυτοί οι άνθρωποι. Αν ήταν ασθενείς θα υπήρχε ένας ιδιαίτερος τρόπος μεταφοράς τους. Και αυτό δεν ισχύει για τα άτομα με αναπηρία, αλλά για τους ανθρώπους που είναι ασθενείς. Υπάρχει ένα πρόβλημα διαθεσιμότητας προσωπικού και κόστους. Αν λέμε ότι θα πρέπει να εξομαλυνθεί η ζωή των ανθρώπων με αναπηρίες δεν μπορούμε να δεχόμαστε αυτά τα εμπόδια. Δεν πρέπει να παραμείνουν, πρέπει να γίνουν αυτά που πρέπει στα αεροδρόμια. Θα πρέπει να δούμε επίσης το πώς εφαρμόζεται ο κανονισμός και θα πρέπει να αναθεωρηθεί και ο κανονισμός. Θα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει με τις αεροπορικές εταιρείες και νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το εξετάσουμε και να το δούμε παντού, αλλά κυρίως με τις low cost υπάρχει το πρόβλημα. Ξέρουμε ότι οι αεροπορικές εταιρείες για να μειώσουν το κόστος θέλουν να προσγειωθούν στο άλλο άκρο του αεροδρομίου ε, με τις δικές τους κάλες ε, για να κατέβει στο αεροπλάνο και να ανέβει στο αεροπλάνο ε, πρέπει να εξασφαλίζει κανείς όχι μόνο την εκτέλεση του κανονισμού αλλά θα και κάνει διακρίσεις ο κανονισμός έναντι των ανθρώπων με αναπηρία. επαναλαμβάνω, αρκεί να δει κανείς τι απαιτούν οι αεροπορικές εταιρείες από το άτομα με αναπηρία για καταλάβει τι γίνεται. Σας ευχαριστώ κύριε που παρουσιάσατε αυτή την αναφορά και θα έχετε την υποστήριξη της σοσιαλιστικής ομάδας ούτω ώστε να κάνουμε όλες τις αναγκαίες ε, μελέτες ούτω ώστε να γίνουν τα απαραίτητα. Σας ευχαριστώ. Θα μιλήσω για την ομάδα του ΕΛΚ, λέει η Πρόεδρος. Εργαζόμαστε μαζί με τη Σολεδάδ όσον αφορά την εφαρμογή της Συμβάσεως των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία και στις μελέτες που διενεργήθησαν σε κάποια κράτη-μέλη διαπιστώσαμε ότι οι καταγγελίες του Σέρμι είναι βάσιμες. Μια αντιπροσωπεία του Σέρμι ήρθε εδώ και κατέθεσε μία από τις αναφορές. Ε, ταυτόχρονα έχουμε και την αναφορά της κυρίας Μαρασαμπάλα, η οποία έζησε στο πετσί τη την κατάσταση. Της απέτησαν να συνοδεύεται. Αυτός ο κανονισμός λοιπόν του 2006 ε, είναι στα όρια όσον αφορά την ερμηνεία που του δίδεται. Ανάλογα με τον πώς ερμηνεύονται τα ζητήματα ασφαλείας και όταν γίνεται η ανάμιξη ασφαλείας και άνεσης πολύ συχνά, ανάλογα λοιπόν με την ερμηνεία ε, απαιτείται από τους ε, ανθρώπους με αναπηρία να συνοδεύονται από κάποιον πληρώντας και το εισιτήριο ή απαιτώντας μία, μάλλον δύο μέρες προειδοποίησης, ε, που αυτό είναι αντίθετο με τη σύμβαση του ΟΗΕ. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει ο κανονισμός να είναι αρκετά σαφής, ούτως ώστε να μην επιτρέπει ερμηνείες ε, και να δημιουργούνται συγχύσει. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σαφέστατο. Δεν είναι τόσο ξεκάθαρο, διότι στην Ισπανία υπήρξαν πάρα πολλέ ε, περιπτώσει τέτοιε. Υπήρξαν πολλέ περιστάσει παρόμοιε το ΣΕΡΜΙ το έλαβε υπόψη αυτό. Υπήρξαν λαθασμένες ερμηνείες του κανονισμού από τι αεροπορικέ εταιρείε όπου έγινε ανάμειξη της άνεσης με την ασφάλεια, παραβιάζοντας έτσι τα δικαιώματα ισότιμης αντιμετωπίσεως των ανθρώπων με αναπηρία εν συγκρίση με τους άλλους ανθρώπους. Εγώ θα κάνω μια πρόταση. Θα μου πείτε τι σκέφτεστε, θα δώσω μετά το λόγο σε εκείνους που θέλουν να μιλήσουν και στους αναφέροντες. Εγώ θα ήθελα αυτή η αναφορά να διαβιβαστεί στην Επιτροπή Μεταφορών, ούτω ώστε η Επιτροπή των Μεταφορών να αξιολογήσει τις δυνατότητες που υπάρχουν, να ζητηθεί μια τροποποίηση του κανονισμού. Θα στείλουμε επίσης στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ τον ανθρώπο με αναπηρία που συνδέεται άμεσα με το ΣΕΡΜΗ την αναφορά αυτή. Και προτείνω εν συνεχεία η Σολεδάδ και εγώ να χρησιμοποιήσουμε όλες τις πληροφορίες που θα συλλέξουμε στο έργο που κάνουμε για την εφαρμογή της συμβάσεως και να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ε, υλοποίηση της ε, συμβάσεως και ποιο βαθμό. Θα δώσω το λόγο τώρα στον ε, αναφέροντα. Α, όχι. Το λόγο στον κύριο Γιάρ. Δεν ναι, θέλω τώρα να επαναλάβω αυτά τα οποία είπε τόσο ωραία η πρόεδρος μας. Μία μικρή διαφορά απόψεων υπήρχε. Μάλλον όχι, θα ξεκινήσω με τα καλά νέα. Όπως είπε η Κομισιόν έχουμε έναν κανονισμό αλλά η ερμηνεία είναι ελαφρώς διαφορετική οπότε πιθανώς θα πρέπει να επανέλθουμε στο θέμα και το θέμα το οποίο βεβαίως είναι ενδιαφέρον είναι πρέπει να αλλάξουμε τον υφιστάμενο κανονισμό ε, ή, ή αρκεί μια νέα ερμηνεία. Εγώ είμαι πρακτικός άνθρωπος. Δεν με ενδιαφέρει τι από τα δύο θα γίνει, αρκεί να βελτιωθεί η κατάσταση για τους ανάπηρους. Και θα πρέπει νομίζω να ε, το στείλουμε και στην αρμόδια επιτροπή και να τους πούμε τι θέλουμε. Όχι να τους πούμε λάβετε υπόψη στην Επιτροπή Μεταφορών, αλλά θέμε αυτό το πράγμα. Και εμένα δεν με ενδιαφέρει, ας παραμείνει ο ίδιος ο κανονισμός και να αλλάξουμε την ερμηνεία. Ή ξέρω εγώ εάν θεωρούμε πως χρειάζεται μία βελτίωση του κανονισμού. Γιατί νομίζω τα, ε, οι εξειδικευμένες επιτροπές θα κάνουν, κάνουν αρκετά καλά τη δουλειά τους. Απλά πρέπει και εμάς να μας πούνε τι θα κάνουν όντως για να γίνει κάτι γιατί κάτι δεν λειτουργεί στην πράξη, στην πρακτική εφαρμογή. Αυτό θέλουμε να αλλάξουμε. Οπότε αυτό σας παρακαλώ στην επιστολή την οποία θα απευθύνουμε. Ευχαριστούμε Πίτερ. Τον λόγο έχει ο αναφέρον. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων που πήραν το λόγο, θα ήθελα να προσθέσω πως δύο πράγματα έχουν ιδιαίτερη σημασία κατά τη γνώμη μου. Η σύμβαση ε, το, του ΟΗΕ είναι ένα νέο στοιχείο για ε, τα ΜΕΑ. Ενώ οι ρυθμίσεις για τις αεροπορικές εταιρείες ε, Ε, υπακούν σε μια διαφορετική λογική. Πρέπει να προσαρμοστούν τα άτομα και όχι το σύστημα στις ανάγκες των ατόμων. Το αντίθετο μοντέλο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με σύμβαση που έχει επικυρωθεί από διάφορα κράτη-μέλη προβλέπει ε, κάλυψη για την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ορισμένα κράτη-μέλη από πλευρά, ε, παραδείγματο χάρη, των αεροπορικών εταιρεών. Μπορεί μια εταιρεία να ε, αρνηθεί την επιβίβαση ή να επιβάλλει την υποχρέωση να υπάρχει συνοδός για το άτομο με αναπηρία. Το αποτέλεσμα ποιο είναι, επιλέγει τους αερομεταφορείς που δεν ε, προβάλλουν αυτά τα κολλήματα το, το άτομο με αναπηρία για να μπορέσει να ρυθμίσει αυτή την προβληματική κατάσταση. Οι ανάπηροι δεν είναι ασθενείς, είναι, ε, η, η αναπηρία είναι μια ε, κατάσταση στην οποία βρίσκεται ένας άνθρωπος και χρειάζεται βοήθεια για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει. Οπότε δεν είναι δυνατόν να ζητείτε να συνοδός, δηλαδή παραβιάζει αυτό από μόνο του τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου, να αναθεωρηθεί ο κανονισμός για να υιοθετηθεί ένα νέο μοντέλο, το οποίο θα είναι ξεκάθαρο για να γνωρίζουν όλοι τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και να μην επαναληφθούν περιπτώσεις όπου κάποιοι παίρνουν αποφάσεις για άλλους μέσω της ε, άρνηση της επιβίβασης, παραδείγματο χάρη. Η άρνηση τη επιβίβαση είναι πραγματική παραβίαση ε, των δικαιωμάτων, διότι δεν υπάρχει κανένας αντικειμενικός λόγος, πρόεδρος. Ωραία, θα στείλουμε με την δέουσα αιτιολόγηση το, την αναφορά σας ε, στην Επιτροπή Μεταφορών. Λέγοντας ότι ε, αμφισβητούμε την ερμηνεία του κανονισμού για να εξεταστεί αν πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισμός, αν πρέπει να εκδοθούν καθηγητήρες γραμμές για την ερμηνεία του κανονισμού. Θα στείλουμε τα σχετικά έγγραφα και στο φόρουμ των ΑΜΕΑ και θα σας ενημερώσουμε για το, τα όσα θα κάνουμε για την εφαρμογή της σύμβασης στο ΙΕ. Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε τον αναφέροντα και περνάμε στο σημείο 11 της ημερήσιας διάταξης Ε, είναι η αναφορά 0617 που θα μας παρουσιάσει ο Ρίτσαρντ Μπάξτον Βρετανικής Ιθαγένειας ε, για τον καταστροφικό και αυτό το αντίκτυπο του υπαίθριου ρηχείου στο Φώση Φράνα θα μας μιλήσει για την υγεία των κατοίκων. Συνοδεύεται από τον συνήγορό του ο αναφέρον. Θα του δώσω το λόγο για να μας εξηγήσει το περιεχόμενο της αναφοράς. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Περιμένω για ένα PowerPoint, να ανάψει το PowerPoint στο κοινό υπολογιστή. Um, uh, Είναι καθυστερή καθυστερεί λίγο, εν πάση περιπτώσει, να σας πω. Γι' αυτό εδώ πέρα πρόκειται για τον αντίκτυπο ενός ε, ανοιχτού ορυχείου, ανθρακορυχείου, στη Φώση Φράν στην ε, Νότια Ουαλία ε, το οποίο απέχει ελάχιστα μέτρα από τα σπίτια στην ε, περιοχή μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είναι η Ουαλία στο χάρτη. Εδώ πέρα έχουμε το Μέρθυρ Τίτφιλ στη Νότια Ουαλία. Και εδώ πέρα έχουμε το χάρτη της ε, περιοχής, ε, ε, βλέπετε τον οικισμό στο κέντρο και το ανοιχτό ανθρακοριχείο είναι εκεί που πέφτουν οι λέξεις Merthyr στο χάρτη. Έτσι έχετε τώρα μία εικόνα της έκτασης. Πρόκειται για 400 εκτάρια. Εκεί βρισκόμαστε λοιπόν Τώρα έχουμε μία εικόνα εδώ πέρα του ανοιχτού ανθρακοριχείου. Δεν είναι ε, μία τρύπα στο έδαφος, είναι ένας λόφος ε, που βρίσκεται πάνω από την πόλη. Και εδώ πέρα έχουμε την άποψη από το ανοιχτό ανθρακοριχείο κοιτώντας τα σπίτια. Τα βασικά σημεία αναφέρονται, 400 εκτάρια έκταση, 11 εκατομμύρια τόνοι άνθρακα έχουν εξορυχθεί σε 15 χρόνια, μιλάμε 36 ε, μέτρα από το κοντινότερο σπίτι, βεβαίως ε, προκαλεί και εκπομπή φυσικών αερίων, ιδιαίτερα μεθανίου, η εξόρυξη και καίγεται μετά ο άνθρακας αυτός στον ε, σταθμό ηλεκτροπαραγωγής του Άμπερθο, ο οποίος επίσης ελέγχεται σε μια διαδικασία επιπαραβάση λόγω των υπερβολικών εκπομπών οξυδίου του αζότου. Πηγαίνει δηλαδή και ε, ο άνθρακας αυτή τη στιγμή σε ένα σταθμό ο οποίος επίσης ελέγχεται και είναι παράνομος. Είχαμε διάφορες διαδικασίες στα δικαστήρια 2005 ήδη οι κάτοικοι προσέφυγαν, ε, απορρίφθηκε η υπόθεση το 2007, 2008 καταθέσαμε μία αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2010 πλέον 5.000 κάτοικοι, 500 κάτοικοι με συγχωρείτε, ζήτησαν από ένα δικαστήριο να σταματήσει την λειτουργία το ανθρακοριχείο. Στην πράξη απολύθηκε γιατί δεν είχαν λεφτά για να πληρώσουν την ε, δικαστική διαδικασία. 2011 η κυρία Όστιν ζήτησε ακριβώς μια, το ευεργέτημα της παινίας για να μπορέσει να καλύψει το κόστος και 24 Δευτέρου του 15 τον προηγούμενο μήνα το ανώτατο δικαστήριο απέριψε το αίτημα της κυρίας Όστιν. Έχουμε λοιπόν και, και παράβαση της ε, οδηγίας 85337 ε, γιατί δεν συμμορφώνεται με τις συνθήκες λειτουργίας. Επίσης δεν αντιμετωπίζονται οι όροι ε, λειτουργίας όσον αφορά τα εργασιακά και βέβαια δεν αντιμετωπίζεται το ζήτημα των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Η σχετική οδηγία λοιπόν λέει πως θα πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένοι όροι όσον αφορά τον θόρυβο και τη σκόνη και εμείς θεωρούμε πως το Ηνωμένο Βασίλειο παραβιάζει την οδηγία για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε σχέση με τις ε, συνθήκες αυτές. Ε, κατόπιν. Ε, ο δεύτερος λόγος για τον οποίο θεωρούν πως είναι παράνομο αυτό το ανθρακοριχείο είναι ότι παραβιάζει τη σύμβαση του Άρχους η οποία επίσης ενσωματώθηκε στην οδηγία για τη μελέτη περιβαλλοντικών ε, επιπτώσεων και άρα θεωρούν πως το Ηνωμένο Βασίλειο παραβιάζει το άρθρο 11 της σχετικής οδηγίας. Και κάτι πιο ουσιαστικό, το τρίτο σημείο, μια παραβίαση της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα τους εξή. Ε, των εξή στόχων της ανάγκης καταπολέμησης του ε, φαινομένου του θερμοκηπίου. Αν υπάρχει ανάγκη τώρα δεν χρειάζεται. Το Ηνωμένο Βασίλειο εξάγει ηλεκτρική ενέργεια. Το συγκεκριμένο εργοστάσιο καύσης το Άμπερθορ επίσης εκπέμπει υπερβολικά πολλούς ρήπους. Οπότε θεωρούμε πως εδώ πέρα παραβιάζεται το άρθρο 191 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν αποζημιώνεται η τοπική κοινότητα και ως συνήθως βεβαίω το Ηνωμένο Βασίλειο προτείνω να σκάψουν και την άλλη μεριά του βουνού για να εξορίξουν άνθρακα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εδώ πέρα έχετε άλλη μια εικόνα της περιοχής μας, άλλη μια φωτογραφία. Σας ευχαριστώ. Δίνουμε τώρα τον λόγο στην ε, Κομισιόν, την κυρία Γκρός. Ερεύνηση Ευρωπαϊκή Επιτροπή ψηρά ετών την αναφορά και στην τελευταία κοινοποίηση θα είδατε όσον αφορά την οδηγία στείλαν πληροφορίες του 2013. Προφανώς μόλις λάβαμε τις συμπληρωματικές πληροφορίες εχθές και συμπληρώνονται περαιτέρω από τον κύριο Στούγκ αυτά που είπε θα δώσω μια απάντηση τώρα, αλλά κάποια θέματα ίσως θα πρέπει να εξεταστούν από όταν θα λάβουμε λεπτομερέστερες ε, πληροφορίες για το όλο υπόβαθρο. Αρκετές, ε, αρκετοί ισχυρισμοί γίνονται, οι περισσότερες αξιολογήσεις που πραγματοποίησαμε δυνάμει της αξιολόγησης επιπτώσεων για το περιβάλλον είναι στις τέσσερις ανακοινώσεις που έχετε μπροστά σας, οπότε δεν θα επαναλάβω τα στοιχεία που περιέχονται σχετικά με το θέμα της πρόσβασης στη δικαιοσύνη, όπως γνωρίζει και ο Στούξ, ερευνήσαμε το θέμα επί καιρών και κινηθήκαμε κατά του Ηνωμένου Βασιλείου κατά παράβαση για υπερβολικό κόστος των διαδικασιών δικαστικής αναθεώρησης. Αυτή η δράση υπήρξε επιτυχής για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρσι, το 2014 με άλλα λόγια, και συζητούμε με τον Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με το πώς δίνουν συνέχεια στο όλο θέμα. Προφανώς θα ενδιαφερόμαστε να δούμε ποια είναι η πρόσφατη απόφαση, η άρνηση του δικαστηρίου να εξετάσει το θέμα και κατά πόσο αυτό εμπίπτει στην οδηγία EIA. Από το έγγραφο που λάβαμε χτες ε, φαίνεται ότι συζητήθηκε το θέμα στα εθνικά δικαστήρια κατά πόσο αυτή η δράση εμπίπτει στην εντολή της ε, αναλύσεως ε, επιπτώσεων και κατά πόσο προσφυγή στο δικαστήριο είναι εκτός του πλαισίου. Η άλλο ισχυρισμό αφορά τον, το σταθμό του Άμπαθορ, παραγωγή ενέργειας. Αυτό είναι ένα θέμα που παρακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για παραβιάσει όσον αφορά εκπομπέ οξυδίων του αζότου. Ε, η γνωμοδότησή μας εξεδόθη το τέλος του περσινού έτους ε, και εξετάζουμε τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν στην όλη διαδικασία αυτή. Τόσο αφορά τις εκπομπέ αερίων του θερμοκηπίου, η αρχική απόφαση περί αυτού ελήφθη υπό την προηγούμενη οδηγία που δεν αναφέρει την αλλαγή του κλίματος σαν θέμα προς ανάλυση, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιέγραψε στην ανακοίνωσή της του 2013 ότι τα έργα του θερμοκηπίου, οι σχετικέ εκπομπέ των αερίων θερμοκηπίου θεωρούνται ότι είναι ένα τμήμα τη κανονική αξιολογήσεω. Προφανώ εδώ δεν αναλύουμε την καύση του καυσίμου. Το έργο, όπω αξιολογεί το σύμφωνο οδηγία, θα αφορούσε την εξόριξη του άνθρακα. Η καύση του καυσίμου δεν θα λαμβανόταν υπόψη από την ανάλυση. Ο άνθρακα μπορεί επιτόπου να καεί στην Ουαλία και αλλού. Αλλά οι κομπέ μεθανίου είναι αέρια του θερμοκηπίου και θα ήταν σχετικό ζήτημα προ ανάλυση. Όσον αφορά την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου, προφανώ ίσω να υπάρχει μια νέα πτυχή και έχουμε αναθεωρημένη οδηγία ΕΕ, η οποία θα αναφέρεται σαφώ στην αλλαγή του κλίματο, που θεωρείται ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη αυτή πτυχή οπότε θα ήταν κάτι εφαρμοστέο από το 2017 αλλά ακόμα και αν η απόφαση λαμβανόταν πριν την θέση ισχύ της νέα οδηγία, νομίζω ότι οι προσανατολισμοί μας είναι αρκετά σαφής ότι οι εκπομπέ αερίων του θερμοκηπίου θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Προφανώς αυτό θα αφορά τη νέα εφαρμογή που εξετάζεται για την επέκταση του πεδίου εφαρμογή. Ευχαριστώ. Πολύ καλά. Υπάρχουν παρεμβάσεις. Απλευρά βουλευτών δεν υπάρχουν παρεμβάσει. Θα δώσουμε το λόγο εκ νέου στον αναφέροντα. Ευχαριστώ Προέδρε. Επανερχόμενο σε αυτά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι εκπομπέ αερίων του θερμοκηπίου πράγματι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στα πλαίσια της εξορυκτικής διαδικασίας η καύση του άνθρακο είναι άμεση συνέπεια της εξόριξης του άνθρακος από ένα ανοιχτό ρηχείο. Οπότε τα σωρευτικά αποτελέσματα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στα πλαίσια της οδηγίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κάλυψε το πρώτο σημείο, δηλαδή τον πρώτο ισχυρισμό ότι υπάρχει παραβίαση της οδηγίας όσον αφορά τη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική δήλωση που εξεπονήθηκε το 2005. Υπήρξε μια περιβαλλοντική ε, ε, ε, δήλωση που εξέδωσε η επιχείρηση του ανοιχτού ρηχείου και είπε ότι θα κάνουμε τα χύψη και ωμέγα ώστε να συμμορφωθούμε με το νομικό πλαίσιο και το ανοιχτό αυτό ρηχείο, ανθρακορυχείο, να μην παράγει χορύπανση και σκόνη. Αυτός ήταν ένας από τους όρους για τους οποίους ε, η εξόριξη ότι θα υπάρχει συμμόρφωση με την περιβαλλοντική επιταγή και λέμε ότι παραβιάζεται. Κατανοώ πλήρω και δέχομαι ότι πρώτερες ανησυχίες που εφήγησαν από την αναφορά εκαλύφθησαν από το Ηνωμένο και κάποια προβλήματα ε, ελήφθηκαν. Αλλά τώρα το 2015 ε, υπάρχει ανησυχία για την πρόσφατη δικαιοσύνη για να προσπαθήσουμε να σταματήσουμε το θόρυβο και τη σκόνη από ένα έργο που αδειοδοτήθηκε σύμφωνα με την οδηγία e IAA και υπάρχει δεύτερη πτυχή, το δεύτερο σημείο σχετικά με τη μη συμμόρφωση με την οδηγία και ότι υπάρχουν όροι που εξακολουθούν να μην πληρούνται όμως από ό,τι φαίνεται μπορεί να χορηγείται άδειο αν πει κανείς ότι θα κάνει τα πάντα για να αποφύγουν τα προβλήματα και μετά αγνοούνται όλα αυτά τη στιγμή που θα πάρει κάποιο την άδεια. Και λέμε ότι αυτό δεν είναι σωστή προσέγγιση όσον αφορά την εφαρμογή τη οδηγία. Και το τρίτο, όσον αφορά την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου, πράγματι είναι γενικότερη ανησυχία και ίσω να μην είναι παράβαση τη οδηγία, αλλά υπό το φω της εκθέσεως του 2012 EAA που έλεγε ότι υπάρχουν σημαντικές ανησυχίες για, την, για τις επιπτώσεις για την αλλαγή του κλίματος στην Ευρώπη και εκτός αυτής υπό το φως ανακοινώσεως της υιοθετήσεως μάλλον του πρωτοκόλου του Παρισιού αρχές του μηνός αυτού στηρίζοντας τη δράση για την αλλαγή του κλίματος φαίνεται ότι δεν είναι ενδεδειγμένο να συνεχιστεί αυτού του είδους η επιχείρηση με το ανοιχτό ορυχείο όταν οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου δείχνουν και λένε ότι πρέπει κατεπηγόντως να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου λόγω των συνεπειών που έχουν για την αλλαγή του κλίματος. Αυτή η πτυχή, δηλαδή η εξόριξη του άνθρακος, η κάψη του άνθρακος επιτόπου και εκπομπές που προκαλούνται, ε, ίσως είναι ένα τέλειο παράδειγμα του πώς να μην καταπολεμείται η αλλαγή του κλίματος. Και θέλω, θα θέλαμε η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο, αυτό να το λάβει υπόψη της, να θεωρηθεί σαν υπόδειγμα αυτή η υπόθεση όπου πρέπει να αναλυφθεί η δράση και δείχνει τα πολύ κακά παραδείγματα ε, που μας δείχνουν αυτά τα ανοιχτά ανθρακοριχεία. Ευχαριστώ. Ο Πίτερ. Αν κατάλαβα καλά την Κομισιόν, είπε πως χρειάζεται πληροφορίες για να αξιολογήσει την κατάσταση. Υποθέτω ότι ξέρετε τι χρειάζεστε. Οπότε προτείνω να κρατήσουμε ανοιχτή την ε, αναφορά αυτή μέχρι να λάβει η Κομισιόν τις ε, πληροφορίες γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να κλείσει και αυτή η αναφορά. Οπότε το, το ερώτημά μου είναι σε πόσο καιρό το βλέπετε, σε πόσους μήνες, κάνα τρίμηνο. Εν πάση περιπτώσει πότε θεωρείτε ότι θα έχετε τις πληροφορίες. Παρακαλώ. Δεν έχουμε ακόμα τις πληροφορίες. Λάβαμε και εμείς χθες ε, την παρουσίαση αυτή με το PowerPoint ε, χθες, ε, αλλά εδώ πέρα διατυπώνονται νέοι ισχυρισμοί και προφανώς απαντάμε σε αυτά τα οποία μας στέλνουν λεπτομερώς, αλλά από το 2013 δεν έχουμε λάβει τίποτα άλλο. Δηλαδή, εγώ ξεπλάγει λίγο από αυτά που είδαμε σήμερα, αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Τώρα υπάρχουν δύο άλλα ζητήματα που έχουν προκύψει. Πρώτα απ' όλα εκρεμεί υπόθεση στα εθνικά δικαστήρια και από ό,τι κατάλαβα από αυτά που μας έστειλαν χθε, το συγκεκριμένο ζήτημα για τους όρους ε, λειτουργίας, που είναι ένα νέο ε, ζήτημα, είναι νέο θέμα και στο ευρωπαϊκό δίκτυο σε σχέση με την οδηγία για, την, ε, για τις επιπτώσεις, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Δηλαδή η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχει στόχο την προαδειοδότηση διαδικασία. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει στα εθνικά δικαστήρια, πώς εξέτασαν το ζήτημα και ποιοι είναι οι όροι τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που ισχυρίζονται εδώ πέρα οι άνθρωποι ότι έχουν παραβιαστεί. Ε, και μέχρι να ξέρω αυτέ τι λεπτομέρειε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση στον αναφέροντα. Για την ε, περίοδο πριν από την ε, ένταξη λειτουργίας του υπεθρίου αυτού ορυχείου. Και θα ήθελα να ξέρω ακριβώς ε, αν υπήρξε μια δημόσια διαβούλευση πρώτον αρχίσει να λειτουργεί το ορυχείο. Γιατί έχουν περάσει 7 χρόνια από τότε που υποβάλλατε την αναφορά. Από ό,τι καταλαβαίνω, 2000, το 2005, δύο χρόνια δηλαδή πρωτού υποβάλλετε την αναφορά, αναλάβατε τις πρώτες δράσεις. Και από ό,τι φαίνεται, παρεμφερείς αναφορές ε, προέρχονται και από όλα μέρη της Ευρώπης. Η επόμενη αναφορά, παραδείγματος χάρη, θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν αν έγιναν δημόσιες διαβουλεύσεις με το δέοντα τρόπο και ποιο ήταν το ε, αποτέλεσμα τους ε, και τα συμπεράσματα που αντλήσατε από τη δημόσια διαβούλευση. Δίνω το λόγο στον αναφέροντα. έγινε μια διαβούλευση προτού να συγκροτηθεί η Επιτροπή μας. Ε, κατά το αναμενόμενο, λαμβάνοντας υπόψη και τις ανησυχίες ε, των ε, περίοικων. Ε, όμως αυτές ε, οι ανησυχίες σχετίζονται με το θόρυβο, την χορύπανση και τη σκόνη. Και ε, μας είπαν ότι καλυπτόμαστε από την περιβαλλοντική δήλωση. Όμως δεν έχει εφαρμοστεί τίποτα και ακριβώς ε, περί αυτού πρόκειται. Γι' αυτό ακριβώς ε, ζητήσαμε να επανέλθει η αναφορά διότι υπάρχει πρόβλημα με αυτήν την περιβαλλοντική δήλωση. Όταν επί τη των πληροφοριών ε, της περιβαλλοντικής δήλωσης ε, του φορέα ε, αγνοούνται ουσιαστικά οι συστάσεις και έχει δοθεί υπόσχεση στους περιοικού ή έχει υπάρξει μια υπόσχεση για ανάληψη δράσης επί τη βάση των συστάσεων της περιβαλλοντικής δήλωσης, τότε τι γίνεται, πρέπει να αναλάβουν οι ίδιοι δράση και τότε προσπαθήσαμε να δράσουμε το 2010 ε, με διάφορα ένδικα μέσα. Η απόπειρα είναι να υπάρξει μια προστασία για το δικαστικό κόστος. Ε, Στο Ηνωμένο Βασιλείο είναι πάρα πολύ υψηλό το δικαστικό κόστος ε, και το Ηνωμένο Βασίλειο έχει κρυθεί ότι δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις σχετικά με το κόστος νομικής διαδικασίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι εξετάζει και άλλα συναφή ζητήματα, μεταξύ των οποίων και αυτό. Όμως δεν σημαίνει ότι είναι σύνομα αυτά που συμβαίνουν επειδή υπάρχει συμμόρφωση με την απόφαση του Δικαστήριου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, του 2014. Υπάρχει σύμβαση του Όρχης που συζητήθηκε για την περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπάρχει μη συμμόρφωση. Διαπιστώθηκε μη συμμόρφωση. Εξακολουθεί να μη συμμορφώνεται εξάλλου με τη Σύμβαση ορχήση το Ηνωμένο Βασίλειο και λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως ότι Λέει μάλλον η Επιτροπή μας ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτε περισσότερο από αυτό και εξακολουθούν να ε, ενοχλούνται από την χορύπανση και τη σκόνη η περίκη. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Σας προτείνω να παραμείνει ε, ανοιχτή η αναφορά και να αναφέρον παρακαλείται να αποστείλει ε, να αποστέλει εφ' εξής όλες τις ε, πληροφορίες ε, στην Επιτροπή μας ε, και θα αποφασίσουμε στο μέλλον. Σημείο 12. Αναφορά 0509 κάθος 2013 της κυρίας Σίλβια Μακοβιάκ εξ του συλλόγου Ναζ Ντόμ για την κατασκευή ε, λίγνη του στην Νότια Πολωνία η ΟΤΑ ε, που εμπλέκονται δεν εκπροσωπούνται αλλά θα πάρει το λόγο η εκπρόσωπος της ΝΑΣ Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σας. Σίλβια Ματσκόβιακ λέγομαι, εκπροσωπώ την Πολωνική Ένωση ΝΑΣ εκπροσωπούμε πάνω από 25.000 ε, άτομα. Στόχο είχαμε να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας ε, κατά της ε, διάνοιξης ενός ανοιχτού λίγνητορυχείου στην περιοχή Διακοπόλσκα. Η άδεια λειτουργίας δόθηκε τον Μάιο του 2011. Εμείς θεωρούμε πως έχουν γίνει κάποια φοβερά λάθη. Παραδείγματος χάρη ε, είχαμε μία διαμαρτυρία την οποία υπέγραψαν 176 ε, άτομα η οποία απορρίφθηκε χωρίς απάντηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και η άδεια λειτουργίας δυστυχώς ε, δόθηκε αλλά βεβαίως είχαμε όπως είπα τραγικά ε, διοικητικά λάθη. Μετά ξεκίνησε βεβαίως η εξόριξη και εδώ πέρα είχαμε πάλι άλλη μια παρανομία και θα έλεγα και παραβίαση των πολιτικών μας ελευθεριών που μας εγγυάται το Σύνταγμα οι ντόπιοι, οι κάτοικοι της περιοχής δηλαδή, ποτέ δεν συμφώνησαν στην εξόριξη. Αλλά μας εξανάγκασαν τα δικαστήρια. Η διαξόριξη άρχισε μόνο με βάση τις αποφάσεις του δικαστηρίου. Οι ντόπιοι εκεί πέρα, οι αγρότες εξαναγκάστηκαν να συμφωνήσουν και παραβιάστηκαν τα δικαιώματά μας. Παρά το ότι η άδεια είχε δοθεί ως προσωρινή, ε, ξεκίνησε αυτομάτως ε, η εξόριξη και παρά το γεγονός ε, πως ε, ε, επρόκειτο για παράνομες ενέργειες εξακολουθεί η εξόρυξη στην περιοχή και από ό,τι φαίνεται θα προσπαθήσει να ανοίξει εντελώς το ανοιχτό αυτό λιγνητό ρηχείο ο επενδυτής και έτσι πολλά χωριά κινδυνεύουν να χάσουν το βιός τους, τα σπίτια τους, τους Μιλάμε για μια περιοχή η οποία είναι πραγματικά ο Σίτο της ε, Πολωνίας. Ε, πολλά δε αγροκτήματα εξυγχρονίστηκαν πρόσφατα με κοινοτικά κονδύλια. Οπότε θεωρούμε πως ε, οποιαδήποτε παρέμβαση σε αυτή την περιοχή είναι προϊόν παρεξήγησης τουλάχιστον αλλά στην πράξη παραβιάζονται εδώ πέρα αστικές ε, ελευθερίες, ε, αλλά και νομοθεσία, υφιστάμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα η οδηγία ε, περί υδάτων. Υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικοί ποταμοί εκεί γύρω και βεβαίως και μια περιοχή Natura 2000 η οποία είναι πάρα πολύ κοντά. Επίσης υποθέτουμε πως ε, παραβιάζεται και ε, οποιαδήποτε αρχή βιώσιμης ε, ανάπτυξης τα ανοιχτά λιγνητορυχεία είναι από τις μεγαλύτερες πηγές εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου και πρέπει να σταματήσουμε αυτά τα σχέδια ενημερώσαμε τις ε, αρχές ε, μεταξύ των οποίων και τον πρόεδρο της ε, Πολωνίας αλλά και τον Υπουργό Περιβάλλοντος. Φτάσαμε στα διοικητικά δικαστήρια και ακόμα περιμένουμε μία απάντηση. Ζητάμε λοιπόν από σας να μας βοηθήσετε να υπερασπιστούμε την πανέμορφη περιοχή μας την οποία βλέπετε εδώ πέρα στις οθόνες και βεβαίως σας προσκαλούμε και να έρθετε εκεί να σας φιλοξενήσουμε για να δείτε και τις λεπτομέρειες της περίπτωσης αυτής. Ευχαριστούμε πολύ την αναφέρουσα. Θα ακούσουμε τώρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Άννα Σαϊκόφσκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σε λίγα λεπτά θα ήθελα να παρουσιάσω πολύ σύντομα τα βασικά στοιχεία της της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον αφορά την κατάσταση. Να αναφέρω εν γέννη ότι πολλά θέματα που θίγονται από την αναφορά φορούν την, ε, την χωροταξία, την χρήση της γης, που είναι ευθύνη και αρμοδιότητα κράτους μέλους στα πλαίσια του περιβαλλοντικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, δηλαδή η οδηγία για την περιβαλλοντική, για την αξιολόγηση αντιχτύπου για το περιβάλλον, χρειάζεται αξιολόγηση ε, των επιπτώσεων πριν δοθεί άδεια. Στην πράξη σημαίνει ότι ο επενδυτής πρέπει να ετοιμάσει μια έκθεση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε όλη τη διαδικασία. Πρέπει να εξεταστούν όλες οι ενδεχόμενες συνέπειες για το περιβάλλον. Να γίνει ιδέως ανάλυση, επίπτωση για επιφανειακά ύδατα, υπόγεια ύδατα, σε γειτονικές περιοχές Natura 2000 ενδεχομένω, στο τοπίο κλπ. Κάτι σημαντικό στην όλη διαδικασία είναι και το εξή. Αφορά και δημόσια διαβούλευση η διαδικασία. Στη δημόσια αυτή διαβούλευση τα ενδιαφερόμενα μέρη θα έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν απόψεις, σχόλια σχετικά με το έργο. Και η διαδικασία κλείνει με απόφαση για τους περιβαλλοντικούς όρους, περιβαλλοντικές συνθήκες. Πού βρισκόμαστε τώρα. Να πούμε σαφώς ότι δεν ξεκίνησε καν η διαδικασία. Ο επενδυτής δεν υπέβαλε αίτηση για την απόκτηση αδείας εκμετάλλευσης. κάνουμε υποθετική αξιολόγηση. Ο επενδυτής απλώς άνοιξε κάποιες τρύπες στην περιοχή, έκανε κάποιες γεωτρήσεις. Άρα, η διαδικασία για την άδεια εκμετάλλευσης δεν ξεκίνησε. Άρα, δεν μπορούμε να διαπιστώσουμε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ενώσης για το περιβάλλον σε αυτή τη φάση. Το ίδιο σχετίζεται και με τις άλλες ανησυχίες. Δηλαδή, αν αυτό το ανοιχτό ρηχείο εγκριθεί ότι θα μειωθεί το ύψος των ε, υπογείων υδάτων και αυτό θα επηρεάσει και την τοποθεσία της Natura 2000 ε, που είναι στα 20 χιλιόμετρα απόσταση. Θα, ε, θα ακολουθούν ίδιες δια, διαδικασίες. Δεν ξεκίνησε η διαδικασία, δεν μπορούμε να συζητήσουμε τον αντίκτυπο για την τοποθεσία Natura 2000 και ούτε παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου. The application to obtain concession to exploit the, uh, the deposits in that area has not been submitted yet. Uh, of course, if the investor applies... Uh, αν επενδύτης κάνει την αίτηση για την εκχώρηση της άδειας, και αν στη διαδικασία για την αδειοδότηση διαπιστωθούν σοβαρές παραβιάσεις, θα κινηθούμε αναλόγως. Bien, gracias. Καλώς. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτά που μας είπατε. Ο κ. Βαλέσο έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αναφέροντες που παρουσίασαν τις απόψεις τους. Είναι πολύ σημαντικό όταν συζητούμε τόσο μεγάλα έργα να λαμβάνουμε υπόψη διάφορες πτυχές και τις θετικές και τις αρνητικές όπως περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ακούσαμε κάποια σημαντικά επιχειρήματα που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από την Επιτροπή μας. Να κατανοήσουμε καταρχάς ότι σχετίζεται το θέμα αυτό με τις πιο σημαντικές γόνιμες περιοχές της Πολωνίας. Γόνιμες για τη γεωργική εκμετάλλευση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι σιτοβολώνας της Πολωνίας. Αυτό είναι το πρώτο επιχείρημα. Δεύτερον, ακούσαμε ότι μέχρι τώρα το Υπουργείο Περιβάλλοντος έδωσε άδεια μόνο για διερεύνηση, για διερευνητικές ε, ε, επιχειρήσεις για την ύπαρξη ε, βοξίτη στην περιοχή. Μέχρι τώρα ανοίχτηκαν 239 τρύπες. Προβλεπόταν 13 ανοίχτηκαν. Από αυτά που μας είπε η αναφέρουσα γνωρίζουμε ότι βάσει των διερευνητικών γεωτρήσεων πιθανότατα θα ζητήσει άδεια επενδυτής για εκμετάλλευση. Σε αυτή τη φάση μπορούμε να συγκεντρωθούμε σε αυτά που μπορούμε να κάνουμε εμείς. Αν κάποιος θέλει να πάρει την άδεια, θα πρέπει να εγκριθούν περιβαλλοντικές πτυχές, θα πρέπει να ανάψει πράσινο φως για την αδειοδότηση. Η Επιτροπή μας λοιπόν θα πρέπει να κάνει το εξής να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη τους φόβους των κατοίκων. Πολύ πιθανόν να υποστεί βλάβη το περιβάλλον. Λοιπόν, εγώ τι λέω, να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Απ' την άλλη βέβαια, να υποβάλουμε και ένα έγγραφο στις πολωνικές αρχές και στο έγγραφο αυτό να συμπεριλάβουμε ανησυχίες όσον αφορά τις διαδικασίες που ακολουθούνται και μετά αποφασίζουμε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα, τι να κάνουμε αργότερα. Πρώτα απ' όλα όμως να ζητήσουμε πληροφορίες από τις πολωνικές αρχές για την πρόοδο των εργασιών, συστάσεις, περιβαλλοντικές αποφάσεις, αλλά και διοικητικές αποφάσεις. Αυτό προτείνω. Να στείλουμε ένα έγγραφο, μια επιστολή στις πολωνικές αρχές και ελπίζουμε να πάρουμε κάποιες απαντήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Βαλέσα. Ο κ. Κούσνιουκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εκ μέρους του κυρίου Βοητσόφσκι που είναι μέλος της ε, Επιτροπής προτείνω να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Δεν θα επαναλάβω τα αναφερθέντα επιχειρήματα αυτά που ακούστηκαν από τους αναφέροντες θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο επενδυτής πραγματοποίησε κάποιες διερευνητικές προσπάθειες. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι είναι αποφασισμένος ο επενδυτής να διαπιστώσει ότι θα ολοκληρωθούν οι όλες οι διεργασίες και θα χορηγηθεί, θα γίνει η επένδυση, θα ολοκληρωθεί. Η αδειοδότηση λοιπόν για τη γεώτρηση χορηγήθηκε για άμεση εφαρμογή. Η τοπική κοινότητα δεν είχε λόγο. Αυτό δείχνει ότι είναι αποφασισμένος επενδυτής να κινηθεί και ότι έχει και επιρροή επενδυτής όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση και ενδεχομένως έχει επιρροή και έναντι των κεντρικών αρχών. Λοιπόν, προτείνω να παραμείνει ανοιχτή αναφορά και ίσως μπορούμε να συμφωνήσουμε με αυτά που είπε ο κ. Βαλένσα, να στείλουμε μια επιστολή, να την αποστείλουμε στις κεντρικές αρχές, να θίξουμε τις ανησυχίες του τόπιου πληθυσμού. Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο. Πρόκειται περί πολύ επίκαιρη συζητήσεως συζητούμε το θέμα πριν ξεκινήσουν οι κατασκευές. Δεν ξέρω, ίσως είναι κάτι αναπόφευκτο, ίσως τελικά να κατασκευαστεί και να αναπτυχθεί αυτό το ρηχείο. Αν θα είναι πολύ αργά τότε και θα συζητούμε το ίδιο θέμα ε, όπως συζητούσαμε και για το θέμα της Ουαλίας όπου ο κόσμος πρέπει να αντιμετωπίσει ήδη τις συνέπειες του ρηχείου που λειτουργεί. Νομίζω ότι αυτό που με εκπλήσει στην όλη αναφορά είναι ότι εκείνοι που υπέβαλαν την αναφορά αισθάνονται αβοήθητοι έναντι ενός μεγάλου επενδυτού, ένας μεγάλος επενδυτής που έχει εμπειρία, πόρους, επιρροή και ξέρουμε ότι ο επενδυτής μπορεί να πλησιάσει τις αρχές. Και εκείνοι που ασχολούνται με τη γεωργία στην περιοχή, που είναι η πιο γόνιμη γη στην Πολωνία, ε, οι άνθρωποι αυτοί αγνοούνται. Και χαίρομαι που τουλάχιστον αυτή η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητούν το θέμα. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, να στείλουμε μια επιστολή, διότι το ότι χορηγείται άδεια για να αρχίσουν γεωτρύψεις ε, αφορά, ίσως σχετίζεται με κάποια υπόσχεση που δόθηκε στον επενδυτή ότι το έργο θα πραγματοποιηθεί. Ίσως υπάρχει κάποιο κενό στην ομοθεσία της Πολωνίας είδος αυτή η άδεια για γεωτρήσεις θα πρέπει να ε, σχετίζεται και με κάποια ε, αξιολόγηση επιπτώσεων. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε να πάρουμε πατήσει από τι πολωνικέ αρχέ και να αφήσουμε και ανοιχτή την αναφορά. Δεν συμφωνώ πλήρω με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Δεν μπορούμε να περιμένουμε. Ίσως αυτή η άδεια για την εκμετάλλευση να δοθεί αυτομάτως. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των πολιτών μας, όχι μόνο όσον αφορά θέματα ιδιοκτησίας, αλλά και το δικαίωμά τους να έχουν κάποια επιρροή, να έχουν λόγο όσον αφορά τη μοίρα της γης τους και του τοπίου τους. Όταν διάβασα την αναφορά σας, είδα ότι πολύ συχνά αναφέρεστε στη χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δυστυχώς αυτή η χάρτα δεν ισχύει στην Πολωνία, διότι η πολωνική κυβέρνηση, οι πολωνικές αρχές δεν συμφώνησαν να συμπεριληφθεί η χάρτα που είναι ένα τμήμα της συνθήκης της Λισαβόνας, δεν συμφώνησαν να εφαρμοστεί αυτή η χάρτα, δεν ισχύει ούτε στην Πολωνία ούτε στο Ηνωμένο Βασίλειο η χάρτα. Όμως έχουμε άλλες οδηγίες στις οποίες θα μπορούσαμε να αναφερθούμε και να προστατεύσουν τα δικαιώματα των πολιτών πρέπει να έχουν λόγο οι πολίτες όσον αφορά το περιβάλλον, τις κοινότητές τους και τα τοπία αυτό θα έπρεπε να αφορά η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Θα πρέπει να κινηθούμε το ταχύτερο δυνατόν, να υποβάλουμε μια επιστολή προ τι κεντρικέ αρχέ τη Πολωνία, αλλά και προ την τοπική αυτοδιοίκηση και να ζητήσουμε την τοπική αυτοδιοίκηση να δώσει κάποιε εξηγήσει. και νομίζω ότι θα πρέπει να αποφύγουμε αυτόματε κινήσει και αυτόματε διαδικασίε. Ευχαριστώ. ευχαριστώ κυρία Νταλή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα ήθελα να εστιάσω σε κάτι διαφορετικό. Ανέφερε κάτι ο αναφέρον, μίλησε για πολιτικές ε, ελευθερίες η κυρία και τόνισε πως αναγκάστηκαν να συμφωνήσουν ε, οι αγρότες. Μα πώς εξαναγκάστηκαν, θα ήθελα να το γνωρίζω αυτό γιατί είναι σημαντικό να ξέρουμε πώς ε, ασκήθηκε αυτή η πίεση. Όταν πήγε μάλιστα το θέμα ενώπιον του ανώτατου δικαστηρίου. Θα ήθελα να γνωρίζω λοιπόν τι έγινε, πότε πήγε ενώπιον του ανώτατου δικαστηρίου για να ξέρουμε και εμείς ε, πόσο, ε, κατά πόσο παρατάθηκε ο χρόνος αυτός και γιατί δεν έχουν ακόμα λάβει απάντηση οι ε, αναφέροντες. Ευχαριστώ κύριο Ζιπ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω δύο ερωτήσεις αν ε, ε, μου επιτρέπετε. Η θέση της ε, τοπικής αυτοδιοίκησης την ε, αρχή ε, της υπόθεσης αυτής είναι το ένα ερώτημα. Και δεύτερον, έχετε κάποιες ε, έρευνες που να αναφέρουν το κοινωνικό κόστος για το ανοιχτό αυτό λιγνητορυχία. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Τον λόγο έχει πάλι αναφέρουσα και αν θέλετε μπορείτε να απαντήσετε και στο ερώτημα της κυρίας Ντάλη. Σας ευχαριστώ. Ματσκόβιακ λέγουμε εγώ, είμαι μέλος της Ένωσης ε, Νασδόμ. Θα ήθελα να συμπληρώσω κάποια πράγματα. και να πω πόσο περήφανοι και ικανοποιημένοι είμαστε για την στάση ορισμένων ε, ευρωβουλευτών που λένε πως ε, η πρόληψη είναι καλύτερη από την ε, θεραπεία. Ο επενδυτής ήταν τυχερός και έπεισε τα δικαστήρια για αυτά τα οποία έλεγε γιατί αναφέρεται σαφώς πως ε, του δίνεται η άδεια για εξόριξη η οποία δεν θα επηρεάζει όμως το δικαίωμα στην ε, ιδιοκτησία. Όμως σαφώς η ε, Γεωργή είναι εναντίον και κατάφερε παραδείγματος χάρη να φέρει την αστυνομία για να επιβάλλει αυτό το οποίο ήθελε. Επίσης έγινε και ένα συνέδριο στο Πανεπιστήμιο του Πόσναν ε, με παρουσία του καθηγητή Ρατάιτεκ και Γκούρσκι και είχαν πει πως ε, η βλάβη του περιβάλλοντος ε, ήταν ε, αναμενόμενη. Τώρα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαίο κάθε κράτος μέλος ε, και η Πολωνία θα πρέπει να μειώσει τις εκπομπές αερίου του θερμοκηπίου. Τι θε, τώρα λοιπόν το ερώτημα τι σχέση έχει με αυτά, ένα λιγνητορυχείο. Επίσης μιλήσαμε για μια περιοχή η οποία είναι ο σιτοπολώνας της Πολωνίας. Ένα τρίτο των τροφίμων ε, της Πολωνίας παράγεται εκεί πέρα. Και οποιαδήποτε ζημιά γίνει θα έχει πάρα πολύ σοβαρές ε, συνέπειες η Κομισιόν ε, μίλησε για διερευνητικές ε, εργασίες ε, ναι αλλά μέχρι στιγμής έχει γίνει ένα 30% των γεωτρησεών και εμείς φοβόμαστε ότι θα θεωρηθεί το μέρος αυτό στρατηγικός πόρος της Πολωνίας και θα υποφέρουμε από αυτή την ε, απόφαση. Θεωρώ πως ε, αυτό το οποίο λέει ο κύριος Βαλέντσα να, να απευθύνουμε μία επιστολή στο Υπουργείο. Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι εδώ πέρα πως θα έκανε υποτίθεται 280 γεωτρήσεις ε, ο επενδυτής και έχει γίνει μόλις το 1 τρίτο μέχρι στιγμής και λέει ο επενδυτής πως ε, υπάρχει πάνω από ένα εκατομμύριο τόνους ε, λιγνίτη εκεί πέρα που μπορεί να εκμεταλλευτεί. Οπότε το σκεπτικό είναι να απευθύνουμε μία επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος ε, για να παρουσιάσουμε τις ανησυχίες μας. Μιλάμε για μια κοινότητα η οποία αντιστέκεται σε έναν επενδυτή. 3.000 άτομα μπλοκάρισαν τον δρόμο, πάνω από 200 τρακτέρ είχαν κλείσει το δρόμο. Διαμαρτυρώμενοι για το άνοιγμα του ανοιχτού αυτού λιντορχείου. Εδώ και τέσσερα χρόνια μας λένε να μην ανησυχούμε και μόνο έρευνες κάνουν, αλλά δεν θα μας ε, ξεγελάσουν, γιατί ξέρουμε πως ε, μόλις βρούνε τον λιγνίτη θα λάβουν και άδεια. Ε, άδεια λειτουργίας και γνωρίζουμε πως ε, η Πολωνία δεν θα έχει κανένα πρόβλημα όσον αφορά παραδείγματο χάρη την ε, παροχή ενέργειας. Τρεις προτεραιότητες υπάρχουν στην Πολωνία. Τα τρόφιμα, η ενέργεια και το νερό. Εμείς ε, θεωρούμε πως η ενέργεια μπορεί να υποκατασταθεί ή να εισαχθεί, αλλά δεν υπάρχει υποκατάστατο για τα τρόφιμα τα οποία παράγονται επί τόπου. Ναι, παρακαλώ. Θα ήθελα να απαντήσω σε κάποιες από τις ε, ερωτήσεις. Ε, τέθη ε, μια ερώτηση που έλεγε πότε έφτασε η υπόθεση αυτή στα διοικητικά δικαστήρια πάνω από ένα χρόνο. Δεν έχω τώρα τον αριθμό της υπόθεσης, αλλά είχαμε πάνω από 167 άτομα τα οποία προσέφυγαν ομαδικά ε, και είχαν προσφύγει και ενώπιον του Πολωνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ε, απευθύναμε και μία επιστολή, δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση από το 2011 ήδη, πριν από τέσσερα χρόνια. Καμία απάντηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Τώρα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για το ενδιαφέρον σας. Ε, ναι, υπάρχουν πάρα πολλά παραθυράκια και πράγματι η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Πρέπει να κάνουμε κάτι τώρα γιατί μετά θα είναι αργά. Και με βάση και την δική μας ε, νομοθεσία. τότε... Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επηρεάσουμε τις αποφάσεις της ε, πολωνικής ε, κυβέρνησης. Οπότε ξέρουμε πως έτσι βεβαίως ε, υπάρχει και το ζήτημα της λυπής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, της οδηγίας για τα ύδατα. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας και ελπίζουμε να γίνουν κάποια συγκεκριμένα βήματα. Ελπίζω λοιπόν να κάνετε κάτι για τους δεκάδες, εκατοντάδες πολίτες που βασίζονται σε σας. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ λέει η Πρόεδρος. Τώρα. Σας προτείνω το εξή. Παραμένει ανοιχτή η αναφορά και θα στείλουμε στις πολωνικές αρχές επιστολή ζητώντα πληροφορίες για αυτό το ζήτημα. Να φέρουμε ότι βρίσκουμε την κατάσταση ανασυχητική. Θα, μόλις ε, έχουμε στη διάθεσή μας ε, τις απαιτούμενες πληροφορίες, τότε θα σας ενημερώσουμε. Τώρα, σημείο 13, αναφορά 0195-2011 του Παουντήλιο Ρος Πράτ. Εξ ονόματος του Καταλανικού Γεωργικού Ινστιτούτου, σαν εισήτρου σχετικά με το έργο του αρδευτικού καναλιού Σεγκάρα Καρή και στη Λέριντα. Ο κύριος ε, ε, Βαντήλιο Ροσπράτη είναι εδώ. Ωραία. Σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. αποτελείται από ε, εταιρείες και από γεωκτήμονες ε, το Καταλληνικό Γεωργικό Ινστιτούτο ε, στην αυτόνομη περιοχή αυτή της Ισπανίας υπάρχει εδώ και 160 χρόνια και έχει ως στόχο την προώθηση της γεωργικής δραστηριότητας. Ε, το 1994 ε, λάβαμε γνώση του, των έργων του Αντευτικού Καναλιού σε Γκάρα Καρίγκες. Ε, είναι ένα κοινοφελές πρόγραμμα και 170 χιλιάδες εκτάρια πλέον θα αρδεύονταν στις πλέον φτωχές περιοχές της ε, καταναλυνικής επαρχίας. Όμως με, την, με το Natura 2000 η αρχική επιφανεία προς άρδευση μειώθηκε πάρα πολύ σημαντικά διότι πάνω από το 40% αυτής της ζώνης βρισκόταν ε, μέσα στις ειδικές περιοχές προστασίας των πτηνών ε, βάση του Natura. Οι γεωργοί λοιπόν που θεωρούσαν ότι θα είχαν νερό ε, προς ε, άρδευση βρέθηκαν αντιμέτωποι με προβλήματα, άρχισαν δημόσιες συζητήσεις και έτσι υπέβαλε το Καταναλικό Γεωργικό Ινστιτούτο αναφορά. Δεν θέλουμε φυσικά να προτείνουμε περιορισμό των προστατευόμενων από το Natura 2000 εκτάσεων, απλώς ζητούμε ε, από ζημιώσεις ε, σε σχέση με τις ε, δαπάνες που έκαναν καταναλυνικές αρχές το 2010 βάσει των περιβαλλοντικών δηλώσεων και έχουμε δύο συγκεκριμένα παραγράφους που είναι πάρα πολύ σημαντικές στην αναφορά. Σε αυτές τις περιοχές που απαγορεύεται η άρδευση θα πρέπει να διεξαχθούν και μελέτες οι οποίες θα αποδίδουν ότι υπάρχει συμμόρφωση ανάμεσα στο πρόγραμμα άρδευση και την προστασία ε, των κοινών, ε, διότι ζητάται συμμόρφωση από τις καταναλωτικές αρχές. Εμεί θεωρούμε ότι ένα μεγάλο μέρος των αποκλειστήσεων περιοχών μπορούν ε, παρόλα αυτά να αρδεύονται και αυτό δεν θέτει σε κίνδυνο την ζωή των πουλιών διότι δεν, αυτό, δεν αποκλείεται από την παρουσία των πτηνών η αρδευόμενη ή μη αρδευόμενη γεωργική εκμετάλλευση, μόνο πρέπει να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των πτηνών. Ε, η ζώνη κοντά στο κανάλι σε Γκαρακαρίκες ε, Έχει γίνει μια μελέτη που αποδεικνύει ότι είναι δυνατόν να ε, υπάρχει άρδευση σε... εχει γινει μια μελετη ταυτόχρονα να βελτιωθούν οι βιότοποι όπου διαβιούν αυτά τα πτηνά. Το ίδιο μπορεί να γίνει και για το ε, κανάλι Σεγκάρα Γκαρίγκα στη Λέριντα. Οι ε, απαιτούμενες επενδύσεις δεν θα πρέπει να γίνουν σε κάποιες από τις ζώνες, ε, διότι η έξοδος από την Ήπεθρο ξύνεται λόγω της έλλειψης επενδύσεων. Εάν δεν μπορούμε όμως, όπως λέει η δήλωση περιβαλλοντικού αντικτύπου, να γίνουν επενδύσεις στην άρδευση, τότε θα πρέπει να δοθούν στις πληγήσεις ε, εκμεταλλεύσεις ε, αποσμιώσεις. Το δευτερεύον σχέδιο που έχει υποβληθεί για τη χρηματοδότηση, ούτως ώστε να ε, γίνει εκτροπή ενός ε, μέρους προς άρδευση ε, κυκισμών που βρίσκονται στα ΠΕΡΙΞ δεν μας βρίσκει αντίθετους όμως πρώτα απ' όλα, προτού ληφθεί μια τέτοια απόφαση, θα πρέπει να διαπιστώσουμε μήπως θα μπορούσε να περιοριστεί η έκταση που αποκλείεται από την άρδευση λόγω του Natura 2000 ουδάλλως, ε, υπονομεύονται οι αρχικοί στόχοι του αρδευτικού κανονίου σε καρακαρίκες. Ευχαριστώ μάλιστα. Ε, μιλήσατε για όλους, εκπροσωπήσατε όλους, ωραία μάλιστα, τότε. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ. Τον λόγο έχει η Κομισιόν. Ο ε, κύριος Σάββατ Μάρτιν είναι εδώ. Είναι εδώ η Κομισιόν. Μάλιστα, ωραία, έχετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Αυτή η αναφορά θέτει δύο ζητήματα σε σχέση με την περιβαλλοντική προστασία. Πρώτον, ο τρόπος με τον οποίο ταξινομούμε τις ε, ζώνες ειδική προστασίας για τα πτηνά και την διαχείριση ή τις δραστηριότητες που ε, μπορούμε να, ε, μπορούν να αναλαμβάνονται μέσα σε αυτές τις ε, ζώνες ειδικής προστασίας. Λοιπόν, το αντικείμενο της αναφοράς εφέρει επί των δύο αυτών ε, ε, τομέων και Δίης έχει καταδικαστεί η Ισπανία από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, διότι δεν έχουν ταξινομηθεί αρκετές περιοχές στη, ως ζώνη, δεν έχουν καταχωριστεί αρκετές περιοχές ως ζώνη Α του προγράμματος Natura και έχει αποφασίσει το δικαστήριο ότι θα έπρεπε να να είναι ζώνη ειδική προστασία σε σχεδόν το σύνολο των εκτάσεων του καναλιού αυτού. Οπότε, αυτές οι δύο αποφάσεις του δικαστηρίου θα πρέπει να εφαρμοστούν από πλευράς των Ισπανικών αρχών. Η ταξινόμηση προβλέπεται στο άρθρο 4,4 της οδηγίας για τα πτηνά και τα κράτη-μέλη πρέπει να ταξινομούν ως προς τον αριθμό ή την έκτασή τους αυτές τις εκτάσεις που προβλέπονται για την προστασία των πτηνών στο παράδειγμα 1 της οδηγίας. Η Ισπανία δεν είχε ταξινομεί σε αυτήν την κατηγορία των ζωνών ειδική προστασία σε αρκετέ περιοχέ. και γι' αυτό καταδικάστηκε από το δικαστήριο η Ισπανία. Κατά την εφαρμογή λοιπόν αυτής της απόφασης η Καταλωνία διεύρυνε, επέκτηνε αυτές τι ζώνε ειδική προστασίας όπω είχαν αρχικά οριοθετηθεί. Υπήρξε λοιπόν επέκταση αυτών των ζωνών. Και Υπάρχει υποχρέωση, όπως είπαμε, καταχώρησης, αλλά υπάρχει υποχρέωση της διαχείρισης αυτών των ε, περιοχών. Αυτό γίνεται από τα κράτη-μέλη, δεν γίνεται από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ταξινόμηση γίνεται επί τη βάση ορνηθολογικών επιστημονικών κριτηρίων και τα κράτη-μέλη προβαίνουν στην ταξινόμηση των περιοχών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το διευκρινίσουμε διότι ο χαρακτηρισμός ε, ζώνη ειδική προστασίας ε, υπάγεται ε, όχι σε οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια ή ασδήποτε φύσης, αλλά σε ορνηθολογικά κριτήρια, όπως σας είπα, ή επιστημονικά κριτήρια. Υπάρχουν βεβαίω άλλα κριτήρια που είναι δυνατόν να συνυπολογιστούν, αλλά όχι κατά την περίοδο της ταξινόμησης ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, εφόσον πρόκειται για μια διοικητική απόφαση, μπορούμε να προσβάλλουμε την, ε, να, να προσβάλλουμε αυτή την απόφαση και θα πρέπει να εξεταστεί αν η Καταλωνία συμμορφούνται με τις ε, διατάξεις που προβλέπονται για την εφαρμογή αυτή τη απόφαση του Δικαστηρίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξετάσαμε λοιπόν το κατά πόσο υπάρχει συμμόρφωση από πλευρά τη καταναλωτική επαρχία και υπάρχει. Σε όλες αυτές τις ε, ζώνες ε, ε, διαβιούν πτηνά που χρήζουν προστασίες βάσει της οδηγίας. Αυτό το κομμάτι έχει σχέση με την ταξινόμηση, αλλά ένα διακριτό ζήτημα είναι η διαχείριση. Η διαχείριση των ζωνών και οι δραστηριότητες που μπορούν να επιτελούνται σε περιοχές ε, του Natura 2000. Αληθεύει ότι υπάρχει και η οδηγία ε, των βιοτόπων, διότι μέσα στο Natura 2000 υπάρχει παραπομπή στο Habitat. Εκεί λοιπόν προβλέπεται μηχανισμός διασφάλισης σε βάση του οποίου οποιαδήποτε προγράμματα δεν ε, συνδέονται με τη διαχείριση και πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο πρώτερης έγκρισης. Ακόμη και αν δεν υπάρχει αρνητικός αντίκτυπος, αν δεν διαπιστωθεί μετά τη μελέτη αρνητικός αντίκτυπος, ε, διαπιστώνεται αν μπορεί ε, να ε, υλοποιηθεί το σχέδιο από την εταιρεία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το σχέδιο αυτό ε, ολοκληρώθηκε, περατώθηκε από την Καταλωνική Επαρχία πριν να εκδοθεί η απόφαση ε, και ε, αποτελείται από δύο σκέλη, από την κατασκευή του ε, καναλιού και από το αρδευτικό πρόγραμμα. Λοιπόν, μετά την απόφαση προβλέπεται διεξαγωγή με, μελέτης περιβαλλοντικού αντικτύπου. Το δικαστήριο Καταδίκασε την Ισπανία διότι ε, προχώρησε σε αυτό το έργο χωρίς να ε, κάνει αυτήν την μελέτη και αυτό που απαιτείται τώρα από την Καταλωνική Επαρχία είναι να ολοκληρώσει το πρόγραμμα χωρίς όμως να πληγούν οι περιοχές, οι ζώνες ειδικής προστασίας και αυτό έγινε από πλευράς Καταλωνίας διότι ε, έγινε μια περιβαλλοντική δήλωση, δήλωση περιβαλλοντικού αντικτύπου μετά από μελέτη για τα προγράμματα υδροδότησης ε, ε, ή για όλα τα υπόλοιπα προγράμματα μετατροπής ε, των βιοτόπων όπου υπάρχουν γεωργικές δραστηριότητες και η καταλονική αρμόδια αρχή, αρμόδια δηλαδή για τη διαχείριση του προγράμματος Natura, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μία σειρά αρνητικών αντικτύπων που ενδεχομένως μπορούν να οδηγήσουν σε καταστροφή των ε, φυσικών χαρακτηριστικών της περιοχής. Όμως, επειδή πρόκειται για ένα κοινοφελές πρόγραμμα εξαιρετικά χρήσιμο, ε, αποφάσισε ε, η κυβέρνηση ότι θα πρέπει σε περίπτωση ζημιών που δεν μπορούσαμε να αποφύγουμε να προβλεφθούν ζημιώσεις. Οι ζημιές που έχουν ε, διαπιστωθεί σχετίζονται ε, με την μετατροπή ενός οικοσυστήματος από ξηρό σε υγρό βιότοπο. Υπάρχει απώλεια τοπίου μετατροπή των εγγενών φυσικών χαρακτηριστικών, παράπλευρες ε, ε, απώλειες και ζημιές που ε, επισύρει το πρόγραμμα άρδευσης. Η περιβαλλοντική δήλωση προβλέπει ότι καλλιέργειες που δεν συνάδουν με τα χαρακτηριστικά της περιοχής και που συνεπάγονται μετατροπή ε, της κυράς σε αρδευόμενη περιοχή δεν πρέπει να επιτρέπονται διότι δεν μπορεί να διορθωθεί ε, η ζημιά που προκαλείται. Αυτά τα διαχειριστικά μέτρα είναι το αποτέλεσμα μιας αξιολόγησης περιβαλλοντικού αντικτύπου ε, και αναφέρονται στη δήλωση περιβαλλοντικού αντικτύπου Ελαμβάνονται υπόψη και στον προσδιορισμό της χρήσης γης του ε, διαχειριστικού σχεδίου. Το διαχειριστικό σχέδιο εγκρίνεται επίση μέσω διοικητική πράξη, μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο προσφυγή ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων. Οπότε, για την περιβαλλοντική διαχείριση, είτε πρόκειται για την ταξινόμηση, είτε για την επανεξιολόγηση, εκ των υστέρων του προγράμματος και την υιοθέτηση με διορθωτικών μέτρων, αντισταθμιστικών μέτρων, ε, καθώς και για τον προσδιορισμό των χρήσεων γης, όλα αυτά ε, έγιναν ε, σύνομα, δηλαδή βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Ευχαριστώ. Από τους βουλευτές συναδέλφους, ποιος θέλει τώρα να μιλήσει, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Βάλτρεντι που είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου για αυτά που μας είπε. Αυτό το κανάλι, το Σεγκάρα Γκαρίγες, κατασκευάστηκε για να μπορεί να μεταμορφωθεί μια ξηρή ζώνη σε ε, γόνιμη ζώνη. Αυτός ήταν ο αρχικός στόχος ε, κατασκευής του καναλιού. Και θα ήθελα να απλώς ότι το μισό της περιοχής που θα πρέπει να αρδευτεί από αυτό το κανάλι είναι μια ζώνη ε, άγωνη. Το πρόγραμμα Natura 2000 αντιπροσώπευε για τους γεωργούς της περιοχής ε, μια ζημιά και θα μπορούσαν να ζητήσουν αποζημίωση οι γεωργοί για αυτή τη ζημιά. Αυτό το κανάλι από τις 8 Οκτωβρίου του 2010 αποτέλεσε αντικείμενο διαφόρων μελετών, κυρίως για τις ειδικέ ζώνες προστασίας των πτηνών, τις περίφημες ΕΠΑ. Ποτέ όμως δεν έγινε καμία εγγύ, ε, μελέτη για να διαπιστωθεί κατά πόσο μπορεί το κανάλι αυτό να κατασκευαστεί και να ταιριάξει με τις ζώνες ειδικής προστασίας των πτηνών. Πώς μπορούμε να πούμε ότι τα δύο έργα είναι ε, παρόμοια. Έχουμε δύο έργα διαφορετικά. Έχουμε το νερό που προέρχεται από το κανάλι Σεγκάρα Γκαρίγες. Αυτό είναι σαφές. Το νερό που προέρχεται λοιπόν από το κανάλι, από το Σεγκάρα Γκαρίγες και πιστεύω ότι η αναφορά θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή για να δούμε αν αυτό το έργο σέβεται όλες τις διατάξεις και αν στόχος της κατασκευής του καναλιού, δηλαδή η άρδευση είναι κάτι πραγματικά χρήσιμο και αν το νερό του καναλιού εν συνεχεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν πόσιμο νερό. Αυτό είναι ένα θέμα, το πρώτο θέμα. Μετά, δεύτερος στόχος είναι ο στόχος της μετατροπής μιας άγονης περιοχής σε αρδευόμενη περιοχή και αυτή η οδευόμενη περιοχή θα περνά από ζώνες προστατευόμενες πτηνών. Αν δεν υπήρχε το κανάλι, η γεωργοί θα ήταν χωρίς νερό. Δηλαδή δεν θα μπορούσαν να καλλιεργούν. Άρα και αυτό είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Και προφανώς θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Ευχαριστώ, δεν ζητάει κανένα άλλο τον λόγο, οπότε μπορεί να ξαναλάβει τον λόγο ο αναφέρον πριν ξανακάνω μια πρόταση. Παρακαλώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ποτέ δεν αμφισβητήσαμε την ταξινόμηση των διαφόρων περιοχών της Natura 2000 θα μπορούσαμε, αλλά δεν το κάναμε ποτέ. Αλλά αυτή η περιβαλλοντική δήλωση του 2010 ποτέ ε, δεν πραγματοποιήθηκε. Δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Λοιπόν, για την ώρα δεν ξέρουμε αν η άρδευση είναι συμβατή με το περιβάλλον ή όχι. Επίσης, υπήρξε μια αναδιάθρωση γεωργική στην περιοχή και αναδιανομή των αγροτεμαχίων και έγινε χωρίς να γνωρίζουμε αν υπήρχε άδεια άρδευσης ή όχι. Αν κάποιοι θεωρούν ότι είναι δυνατόν ταυτόχρονα να γίνει άρδευση και να υπάρχει και προστασία των πτηνών, είναι καλό. Αυτό θέλουμε να ξέρουμε. Μπορούμε να έχουμε ταυτόχρονα και άρδευση και προστασία των πτηνών. Διότι δεν θα ευνοήσουμε μία ζώνη εις βάρος άλλης. Να αρνηθούμε την άδεια της άρδευσης αν εμποδίζει δημιουργεί προβλήματα για όλη την περιοχή. Άρα δεν αμφισβητούμε τις περιοχές ειδική προστασίας των πτηνών που προβλέπονται από την οδηγία Natura 2000. Αυτό που θέλουμε είναι μια πραγματική αξιολόγηση περιβαλλοντικών αντικτύπων να δούμε σε ποιο βαθμό είναι δυνατόν να έχουμε ταυτόχρονα και άρδευση και προστασία των πτηνών. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ που ήρθατε εδώ πέρα και σας ευχαριστώ και για την παρουσίαση που κάνατε. Σημείωσα εδώ πέρα τα όσα είπατε. Ίσως να μην υπήρξε στο παρελθόν διάλογος μεταξύ Κομισιών και Περιφέρειας γιατί είναι πραγματικά ατυχές ε, το πώς κορυφώθηκε αυτή η κρίση. Πρώτο συμπέρασμα λοιπόν θα παραμείνει ανοιχτή η αναφορά αυτή και δεύτερον το θέμα είναι θέμα αρχής, ε, το είπε πολύ σωστά και ο ε, αναφέρον ε, μεταξύ της δραστηριότητα αυτής και της προστασίας ε, του ύδατος και βεβαίως θα δούμε το τι θα γίνει αν υπάρχει αυτή η συμβατότητα και το θέμα είναι ποιο ακριβώς ήταν το πρόβλημα εδώ πέρα και τρίτον και εξίσου σημαντικό το θέμα ακριβώς του συμβιβασμού, ότι προσπαθούμε δηλαδή να αντισταθμίσουμε κάποιες ε, παρεμβάσεις ε, για να δούμε τι ακριβώς ε, προβλέπεται εδώ πέρα. Όλα αυτά πάντα σε συνεννόηση με την Κομισιόν. Θέλουμε λοιπόν, δεν θέλουμε να διαλύσουμε την περιοχή αυτή της ε, προστασίας ε, και όχι όμως ταυτόχρονα ε, να καταργήσουμε και την οικονομική ανάπτυξη. Γι' αυτό ακριβώς παραμένει ανοιχτή αυτή η υπόθεση. Θα απευθύνουμε μια επιστολή στις αρχές. Αυτά λοιπόν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ που ήρθατε και περνάμε τώρα στην επόμενη αναφορά ακόμη μια ισπανική ε, του κύριου Κριστομπάλ Αγκουαδαλάζα εξ ονόματος ε, της Ένωσης Ζωσιασιών ε, Βαλενσιάνα για τις ασθένειες των φυτών. Είναι παρόντες εδώ πέρα οι αναφέροντες. Ωραία, ευχαριστώ. Θα δώσω λοιπόν πρώτα απ' όλα τον ε, λόγο στον κύριο Κριστομπάλα Γκουάσα για πέντε λεπτά για να μας παρουσιάσει την υπόθεση. Έχετε το λόγο. Ε, Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να έρθω και να μιλήσω στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξ ονόματος του Γεωργικού Συνεταιρισμού της Βαλένθια. Ο τομέας των απορροκυπευτικών αντιμετωπίζει τώρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Έχουμε λίγα φυτογενομικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υποφέρουμε από προβλήματα οικονομικά που οφείλονται στην ε, χαλαρότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δίνει πολλές άδειε σε τρίτες χώρες ούτως ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν φυτογενομικές ουσίες που απαγορεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο θα θέλαμε να θίξουμε εδώ σήμερα. Πρόκειται περί πραγματικού προβλήματος για την ε, υγεία των φυτών μας. Το πρόβλημα που δημιουργείται από τις εισαγωγές ε, προϊόντων από τρίτες χώρες. Η παρούσα νομοθεσία δεν είναι αρκετά αποτελεσματική όσον αφορά τους ελέγχους και τις ε, επιθεωρήσεις. Πρόκειται για κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Έχουμε πολλές περιπτώσεις ε, σημαδιών λεκέδων μελανών που βρίσκουμε στα απορροκυπευτικά που ε, εισάγονται από την Νότια Αφρική και προορίζονται για τις ευρωπαϊκές αγορές. Ανάμεσα στο 2010 και το 2014 εντοπίστηκαν μαύροι λεκέδες στα απορροκυπευτικά προϊόντα της Νότιας Αφρικής, δηλαδή 35% από τα απορροκυπευτικά προϊόντα. Ε, είναι απαράδεκτο ποσοστό αυτό. Επίσης, είναι σκανδαλώδες να διαπιστώνει κανείς ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας αντιμετωπίζει με συγκατάβαση, μεγάλη συγκατάβαση και με καχυποψία, ενώ τα προβλήματα που καταγγέλουμε είναι σοβαρότατα, πραγματικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνήθηκε να θεσπίσει μέτρα κατά της Νοτιού Αφρικής, ακόμα και σε περίπτωση εντοπισμού πολλών προβλημάτων όσον αφορά τα προϊόντα που εισήγονται από εκεί καθορίστηκε στο 5 το χρόνο το όριο και τον Οκτώβριο ήδη είχαμε εντοπίσει 28 περιπτώσεις τέτοιες. Οι κοινοτικέ αρχές δεν σέβονται λοιπόν τις υποχρεώσεις τους ενώ είχαν δώσει το λόγο τους στον τομέα μας, στον κλάδο μας και εξακολουθούμε να κατακλυζόμεθα από πορτοκάλια, από μανταρίνια, ε, από την Νότια Αφρική με μαύρους λεκέδες ενώ πρόκειται με πολύ σοβαρή ασθένεια που θα πρέπει να μπει σε καραντίνα τα προϊόντα, πρέπει να μπουν σε καραντίνα, διότι υπάρχει κίνδυνος ε, μόλυνσης ε, που το καταγγέλει και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφαλείας των Τροφίμων. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν ε, απαράδεκτη. Και αυτό που είναι ακόμα πιο ε, ανησυχητικό είναι ότι καταγγέλουμε αυτά τα γεγονότα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η Ισπανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιταλία, η Ελλάδα, όλες οι χώρες που παράγουν στην Ευρώπη προκευτικά τέτοια προϊόντα θεωρούν ότι δεν είναι πρόβλημα ανταγωνισμού, δεν μιλάμε για εμπορικούς φραγμούς, διότι εμείς παράγουμε συμπληρωματικά προϊόντα. Το λέω παρευθείς σε εκείνους που θεωρούσαν ότι πρόκειται περί εμπορικού φραγμού και αθέμητο ανταγωνισμού. Δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Τα προϊόντα μας είναι συμπληρωματικά διότι είμαστε στο βόρειο ημισφαίριο και αυτή είναι στο νότιο ημισφαίριο. Στην απόφαση της 17ης ε, Δεκεμβρίου του 2014 ε, επετράπη να μπουν στην Ευρώπη τουλάχιστον 9 νέες ασθένειες. Άρα μία νέα ασθένεια που εισάγεται στην Ευρώπη κάθε 7 μήνες με όλους τους περιορισμούς που έχουμε όσον αφορά τα φυτογενομικά προϊόντα στην Ευρώπη. Φανταστείτε σε τι κατάσταση θα βρισκόμαστε. Στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρονται μόνο οι οργανισμοί που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση των ελόγου ασθενειών. Όμως δεν αναφέρονται όλες οι ασθένειες. Διάφορες ασθένειες δεν αναφέρονται υπάρχει μία ε, προσθήκη ασθενειών που εισέρχονται, ε, που πλήττουν τα φυτά, με αντίκτυπο τεράστιο οικονομικό για τον κλάδο μας. Αυτή η ατυχής ε, ιστορία είχε δραματικές και άκρως ανησυχητικές συνέπειες τον περασμένο Αύγουστο. εντοπίστηκε αφρικανική μύγα στη, Γαλλικία. Βρήκαμε προηγουμένως και στην περιοχή του Πορτό, του Πόρτο μάλλον, στην Πορτογαλία. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε να εμφανίζεται αυτό το έντομο, η Αφρικανική μύγα, στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Εδώ και 1,5 χρόνο ήδη είχαμε υπενθυμίσει στις εθνικές μας αρχές, αλλά και στις ευρωπαϊκές αρχές, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι θα έπρεπε να ξεκινήσει μεγάλη επιχείρηση πρόληψης και επαγρύπνησης. 1,5 χρόνο μετά Έχουμε το παράσιτο αυτό στην Ευρώπη όπως το είχαμε προβλέψει. Με συνέπειες σοβαρότατες, διότι είναι ένα έντομο που είναι φορέας θανατηφόρων ασθενειών για τα προϊόντα μας. Καταστροφικών ασθενειών. Αυτές οι ασθένειες προέρχονται από ένα βακτηρίδιο, όπως τη Μπακτέρ, που υπάρχει στην Ασία, την Αφρική, στην Αμερική και στην Οκεανία αλλά που δεν υπήρχε στην Ευρώπη. Στη Φλόριντα, στην ΙΠΑ καταστράφηκαν πολλά εκτάρια. Μειώθηκε η, παραγωγή κατά 11%. Ε, στη Βραζιλία 24 εκατομμύρια δέντρα ε, καταστράφηκαν σε ελάχιστο χρόνο. Οπότε για τον ευρωπαϊκό πληθυσμό, για όλες τις οργανώσεις ε, προστασίας των φυτών, ε, πρέπει να κινηθούν κατά της ασθένειας που μπορεί να αποδεκατήσει και τις ε, καλλιέργειες της μεσογειακές. Αυτή η ασθένεια μπορεί να καταδικάσει σε θάνατο όλες τις καλλιέργειες ε, των προϊόντων αυτών, των εσπεριδοειδών στην Ευρώπη και των αποκευτικών. Πρέπει να κινηθούμε να αποφύγουμε την καταστροφή και γι' αυτό κύριε Πρόεδρε στεφόμαστε προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ούτως ώστε να απευθύνει άμεσα έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτως ώστε να επιληφθεί επιτέλους επί του σοβαρότατου αυτού ζητήματος με επαρκή χρηματοδότηση για να χρηματοδοτηθούν τα προληπτικά μέτρα που απαιτούνται και όλα τα αναγκαία θεραπευτικά μέτρα για να εκριζωθεί αυτή, ε, αυτός ο φορέας των ασθενειών από την Ισπανία και την Πορτογαλία. Όσον αφορά το σχέδιο οδηγίας για τα φυτογειονομικά, είναι απαραίτητο να έχουμε ένα νέο κανονισμό που θα προβλέπει αυστηρότερους, πολύ αυστηρότερους ελέγχους τώρα σε σημεία εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση των απορροκευτικών που προέρχονται από τρίτες ε, χώρες. Από τη ΣΥΠΑ, η Ιαπωνία, Κορέα, ή μάλλον αυτές οι χώρες έχουν πολύ αυστηρά καθεστώτα, έχουν δικούς τους επιθεωρητές που πηγαίνουν στις χώρες προέλευσης πριν καν καταφτάσουν τα προϊόντα στα λιμάνια τους, ούτως ώστε επιτόπου ε, να ελέγχεται η υγεία ε, των προϊόντων, εάν ανταποκρίνουν τις προδιαγραφές ή όχι. Ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να εμπνευστεί από αυτή την προσέγγιση των ελέγχων, των επιθεωρήσεων στις χώρες προέλευσης των προϊόντων, όχι για όλες τις εξαγωγές, αλλά εξαγωγές όπως αυτές που προέρχονται από την Νότια Αφρική, που έδειξαν ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Στη νέα οδηγία λοιπόν ζητούμε να υπάρχει ένας θετικός κατάλογος, δηλαδή ένας μηχανισμός που ήδη χρησιμοποιείται για τα ζώα και για τα γιόμιλα, να υπάρχει θετικός κατάλογος χωρών που παρέχουν όλα τα αναγκαία εχέγγυα, ούτω ώστε η παραγωγή να έρχεται με σωστό τρόπο στην ευρωπαϊκή αγορά. Οι χώρες που δεν είναι στο θετικό κατάλογο θα πρέπει να ελέγχονται με πολύ αυστηρότερο τρόπο. Ιδού, αυτό ζητάμε Λυπούμε κύριε Πρόεδρε, για μας τους γεωργούς είναι πάντα δύσκολο να μπαίνουμε σε νομικές διαδικασίες και να στρεφόμαστε κατά των θεσμών, αλλά με μεγάλη ελπίδα στρεφόμαστε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτω ώστε να ζητήσουμε να μας βοηθήσει να βρούμε λύση για να προστατεύσουμε την Ευρωπαϊκή Γεωργία. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας άφησα να μιλήσετε και λίγο παραπάνω για να παρουσιάσετε όλες τις πτυχές ε, της ε, υπόθεσής σας και επειδή είναι τόσο περίπλοκη η υπόθεση έχουμε εδώ πέρα κάποιους από την Κομισιόν, δύο άτομα μάλιστα που θα μιλήσουν. Πρώτα απ' όλα ο κύριος Βόφκαν Καράινχαρτ. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα περιοριστώ εγώ στην πτυχή η οποία αναφέρθηκε πρώτη. Δηλαδή τις ανοχές εισαγωγών. Θα ήθελα να πω το εξής, γιατί ακριβώς είναι σαφές ως προς αυτό το ζήτημα πως εάν ακολουθήσουμε αυτό το οποίο λέγεται εδώ πέρα θα έχουμε παραβεί τις διεθνείς μας υποχρεώσεις και του κανόνες ε, του ΠΟΕ γιατί ε, έχουμε κάνει κάποιες συμφωνίες για υγειονομικά και φυτοϊγειονομικά μέτρα και υπάρχουν άρα κάποιες άνοχες ε, παραδείγματος χάρη το 0,1 για το επίπεδο προσοχής ε, στο οποίο μπορεί κάποιος ε, ετών να αποδείξει ότι ένα υψηλότερο επίπεδο δεν προκαλεί ανησυχίες για τους καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε ε, τα χέρια μας είναι δεμένα. Και τώρα θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον συνάδελφο γιατί η πτυχή των φυτογενομικών μέτρων είναι σαφώς ε, μεγαλύτερη. Ε, μάλιστα. Ο κύριος Καραμίτσιος είναι εδώ πέρα στον κατάλογο μου. Το είπα σωστό, έχετε το λόγο. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. επί της αρχής εμείς ε, συμφωνούμε πως ε, τα μέτρα και οι έλεγχοι πρέπει να ενισχυθούν όλο το σύστημα πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματικό αυτή η αρχή αντανακλάται σε δύο επίπεδα πρώτα απ' όλα στο επίπεδο υιοθέτηση ε, μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεκριμένα αγαθά, για συγκεκριμένα ζυζάνια από συγκεκριμένη προέλευση. Παραδείγματο χάρη αυτό το οποίο αναφέρατε για τα εσπεριδοειδή από την Νότιο Αφρική. Το δεύτερο αφορά τους γενικούς κανόνες που έχουμε για τα προστατευτικά μέτρα για το γενικότερο καθεστώς εισαγωγής για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα από τρίτες ε, χώρες. Θα θέλαμε πρώτα απ' όλα να τονίσουμε πως πέρσι υιοθετήσαμε μάλλον την αυστηρότερη απόφαση ε, για τις αγωγές, η 2014 κάθετος 422 ε, για την εισαγωγή προϊόντων φυτικής προέλευσης από την Νότια Αφρική, αυτή την οποία αναφέρατε και εσείς. Αυτή από το τέλος Ιουλίου άρχισε να ισχύει ήταν το μέσον της σεζόν εισαγωγής αγροτικών προϊόντων από την Νότιο Αφρική. Περιλάμβανε όλα τα πιθανά μέτρα που αφορούν τις ε, εισαγωγές ε, μεταξύ των οποίων ε, και απέτηση για προέλευση από μέρος χωρίς ζυζάνια, δειγματοληψία από το σημείο της παραγωγής, ε, ίχνη λασιμότητα, εντατικοποιημένη έλεγχη πρώτης εξαγωγής και εντατικοποιημένη έλεγχη μετά την εισαγωγή στην επικράτεια της Ένωσης, πάρα πολύ αυστηρή όροι που ισχύουν για την Νότια Αφρική και στα λιμάνια εισόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα είναι ότι οι αφρικανικές αρχές συνειδητοποίησαν ότι δεν μπορούσαν να συμμορφωθούν εγκαίρως. Είχαμε νομίζω πέντε ε, φορτία τα οποία σταμάτησαν λίγες εβδομάδες μετά την εισαγωγή και μετά αποφάσισαν οι νοτιοαφρικανικές αρχές από μόνες τους να απαγορεύσουν την εξαγωγή στην ε, Ευρώπη. Οπότε δεν είχαμε μετά άλλες ανασχέσεις ε, φορτίων. Φέτος θα δούμε την εξέλιξη του καθεστώτος. Φέτος θα έχουμε για πρώτη φορά την εφαρμογή της νέας απόφασης για ολόκληρο τον κύκλο της παραγωγής στην Νότιο Αφρική. Οπότε φέτος θα δούμε τι γίνεται πραγματικά και βεβαίως ανάλογα με την εξέλιξη των ζυζανίων και των ασθενειών θα δούμε αν θα γίνουν πιο αυστηροί οι όροι ή αν θα συνεχίσει η απόφαση αυτή να ισχύει όσο έχει και αυτό είναι σύμφωνο με τις διεθνείς μας υποχρεώσεις γιατί οποιοδήποτε περιορισμοί πρέπει να βασίζονται σε αξιολόγηση κινδύνου και να εφαρμοστούν με μέτρα αναλογικά και αποτελεσματικά μέτρα διαχείρισης του κινδύνου. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, όταν μιλάμε για την πρότασή μας για ε, ένα νέο φυτογεωνομικό κανονισμό, η ίδια η πρόταση αυτή εισάγει ένα αυστηρότερο καθεστώς υπάρχει δυνατότητα προληπτικών προσωρινών μέτρων καταγνώστων κινδύνων. Η προσέγγιση αυτή έχει εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ολομέλεια της 15ης Απριλίου πέρσι και μάλιστα με αυστηρότερους κανόνες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή τη στιγμή η πρόταση αυτή συζητιέται από το Συμβούλιο. Ελπίζουμε ότι η επιλετονικής Προεδρίας το Συμβούλιο θα δώσει μια έντολη για ε, τριμερή διάλογο, διαπραγματεύσει με Κομισιόν και Κοινοβούλιο. Στο Συμβούλιο υπάρχουν επίσης αποκλίνουσες απόψεις για το επίπεδο αυστηρότητας ε, των μέτρων εισαγωγής ε, αυτών. Ελπίζουμε να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση. Τέλος, θα ήθελα να κλείσω λέγοντας πως πρέπει να επανεξετάσουμε τα γενικότερα μέτρα για την εισαγωγή σπεριδοειδών όχι μόνο από την Νότια Αφρική αλλά και από όλες τις άλλες τρίτες χώρες τη Βραζιλία, Αργεντινή κτλ. Οπότε μια τεχνική συζήτηση θα ξεκινήσει σύντομα στο επίπεδο μόνιμης ε, Επιτροπής ε, Ζώων Φυτών Ζωοτροφών και τροφίμων για να καταλήξουμε στις πιο αποτελεσματικές απαιτήσει ε, εισαγωγής για τα εσπεριδοειδή. Μπορώ να σας πω και άλλα, αλλά καταλαβαίνω ότι ο χρόνος πιέζει. Έχω και άλλα παραδείγματα, αλλά είμαστε στη διάθεσή σας. Αν θέλετε τίποτα άλλο, ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Κομισιόν. Ο κύριος ε, Μίσος ε, ζήτησε τον λόγο και μετά θα τοποθετηθώ και εγώ ως βουλευτής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Ισπανική Αντιπροσωπεία του ΕΛΚΑ υποστηρίζει τον αναφέροντα και ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι αποτελεσματικότερη για τους ελέγχους των εισαγωγών από τρίτες χώρες. Θα πρέπει να είναι πολύ αυστηρότερη η έλεγχη και να μην διστάζουμε να λαμβάνουμε στερότερα μέτρα για να προστατευτούν οι ευρωπαϊκές καλλιέργειες. Εγώ είμαι και μέλος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι στα πλαίσια του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου υπάρχουν κανόνες που δύσκολα μπορούν ε, να εφαρμοστούν για την προστασία των καλλιεργειών. όμω καταλαβαίνετε ότι οι γεωργοί δυσκολεύονται να καταλάβουν για ποιο λόγο έχει έτσι η κατάσταση διότι καλό το διεθνέ εμπόριο, αλλά θα πρέπει να, υπάρχουν, θα πρέπει να υπάρχουν και ισότιμοι όροι ανταγωνισμού. Η οδηγία λοιπόν θα πρέπει να διέπει τις εισαγωγές των επιβλαβών οργανισμών, αλλά είναι απαρχιωμένο το περιεχόμενο της με τους νέους κανόνες, θα χρειαζόμαστε ένα νέο κανονισμό. Το σχέδιο εξετάζεται αυτή τη στιγμή από το Συμβούλιο και από το Κοινοβούλιο εξάλλου. Λοιπόν, η πρόταση προσδιορίζει τις ελάχιστες διατάξεις για την εισαγωγή στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης ε, των ελαχίστων προτύπων των προϊόντων, ε, καθώς και τα μέτρα που μπορεί να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να παρεμποδίσει την είσοδο αυτών των προϊόντων. Θα πρέπει με ταχύτητα να κινείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το που διαπιστώνεται η ύπαρξη φυτογενομικού προβλήματος θα πρέπει αμελητή να δρούμε διότι στο παρελθόν παραδείγματος χάρη είχαμε πολλές ε, ειδοποιήσεις ε, ε, αλλά δεν έλαβε κανένα μέτρο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η μαύρη κοιλίδα που μας απασχολεί τώρα έχει οδηγήσει σε πάρα πολύ μεγάλες ζημιές για τους γεργούς. Στα πλαίσια του πρασινίσματος θα πρέπει εμείς να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει ποια μέτρα θα ε, αναλάβει για να αναχαιτήσει αυτή την ε, ασθένεια. Ευχαριστώ. Τώρα θα τοποθετηθώ και εγώ ως βουλευτής και μέλος της Επιτροπής Γεωργικών Υποθέσεων, αλλά βεβαίως και αυτής εδώ πέρα. Το πρόβλημα είναι πολυεπίπεδο. Πρώτα απ' όλα γιατί έχουμε διεθνές εμπόριο και πάντα βεβαίως ε, είναι πρόβλημα για τους Ευρωπαίους γεωργούς όταν έρχονται εδώ πέρα τρόφιμα, φρούτα ε, ή άλλα τέτοια προϊόντα που είναι σε διαφορετικό επίπεδο από αυτά τα οποία ε, εισάγονται εδώ πέρα και είναι σε διαφορετικό επίπεδο από τα εντόπια προϊόντα και είναι βεβαίως και στρέβλωση του ανταγωνισμού αλλά και κίνδυνος για μετάδοση ασθενειών. Οπότε πρέπει να βρούμε έναν μηχανισμό πραγματικά να αντιμετωπίσουμε το σύστημα εντατικά χωρίς ε, βεβαίως να σταματήσουμε το εμπόριο. Αλλά πρέπει να είναι κάτι το αποτελεσματικό. Και βεβαίως χρειαζόμαστε αυτά τα μέσα ακριβώς γιατί όταν μιλάμε για φυτογειονομικά ζητήματα είμαστε πάρα πολύ αυστηροί στην Ευρώπη. Και υπάρχουν ε, βεβαίως ε, και ασθένειες ή ζυζάνια τα οποία εμφανίζονται εδώ πέρα και δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε μετά γιατί δεν έχουμε εγκρίνει ή δεν επιτρέπονται τα αντίστοιχα φυτοφάρμακα. Οπότε νομίζω πως ε, η Κομισιόν το είπε, χρειάζεται εδώ πέρα μία αξιολόγηση αντικτύπου γιατί έχουμε απαγορεύσει κάποια μέτρα φυτοπροστασίας αλλά πάντα ε, στα ψηλά γράμματα αναφέρουμε πως πρέπει να γίνει μία αξιολόγηση αντικτύπου. Δηλαδή αν απαγορεύσουμε μια δραστική ουσία και μετά επανεμφανιστεί μια ασθένεια, ίσως πρέπει να ξαναδούμε την ε, κατάσταση. Εσείς έχετε αυτό το πρόβλημα, ίσως κάπου αλλού στην κεντρική Ευρώπη να έχει εμφανιστεί ένα άλλο ζήτημα, μια δραστική ουσία για την οποία δεν υπάρχει υποκατάστατο. Και το είπε νομίζω η Κομισιόν ήδη πως είναι αρκετά περιοριστικό το Κοινοβούλιο. Εμείς είμαστε στο πλευρό σας και λέμε πάντα πως πρέπει με τα εισαγόμενα τρόφιμα να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί να έχουμε μια δίκαιη δηλαδή αντιμετώπιση και βεβαίως ε, και να τηρούμε ε, και τις προδιαγραφές ε, της παραγωγής. Τα άκουσα αυτό το οποίο η χρειάζεται εδώ πέρα περισσότερη έλεγχη για να λάβουμε και τα σχετικά μέτρα. Τώρα, συνεχίζουμε στην διαδικασία. Τον λόγο έχει πάλι ο αναφέρον και μετά θα συνοψίσω εγώ αλλά όπως είπαμε η αναφορά σας ε, θα πρέπει να γίνει και στην Επιτροπή Γεωργίας. Γιατί ακριβώς ε, είναι πολλά τα ζητήματα, είναι και στρέβλωση του ανταγωνισμού, είναι η φυτοπροστασία. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικά τα ζητήματα και σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ πέρα. Λοιπόν, έχετε τον λόγο και μετά θα συνοψίσω ως πρόεδρος. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την ε, προσέγγιση αυτή που υιοθετείτε, διότι το πρόβλημα αυτό αφορά ολόκληρο τον τομέα το, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε με ελάχιστα μέσα φυτοπροστασίας να αντιμετωπίσουμε ασθένειες που προκύπτουν κάθε 7 μήνες, ε, παραδείγματος χάρη. Ε, με τις εισαγωγές των προϊόντων έχουμε τις ασθένειες ολόκληρο του κόσμου. ενώ σε άλλες περιοχές έχουν μόνο τις δικές τους ε, ασθένειες. Ε, είμαστε σε δυσμενή θέση. Μάλιστα, προτείνω το εξή. Πρώτα απ' όλα παραμένει ανοιχτή η αναφορά και θα πρέπει να την αποστείλουμε και στην Επιτροπή Γεωργίας και παρακαλώ τη Γραμματεία όχι να τη στείλουμε. Θέλουμε γνωμοδότηση από την Επιτροπή Γεωργίας για το θέμα αυτό. Γιατί ξέρω πως μας απασχολεί και εκεί πέρα το ζήτημα. Και, τη... και η σχέση με το διεθνές εμπόριο είναι ένα πρόβλημα το οποίο αφορά και την εμπορική στρατηγική και διάφορα άλλα τέτοια ζητήματα. Οπότε πρέπει να το δουν οι αρμόδιες ε, επιτροπές. Ε, σας ευχαριστώ λοιπόν ακόμη μια φορά και όπως σας είπα είμαστε στο πλευρό σας ε, σε αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, περνάμε άρα στην επόμενη αναφορά. την οποία έχει καταθέσει η Μερέη Γκρός Χάνς εξ ονόματος καθηγητών βιοχημίας μεταξύ των οποίων νομπελίστες και άλλα 140 άτομα σχετικά με την απαλλαγή των μυγών των καρπών από κτηνιατρικούς ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα βάσης οδηγίας 91 4, 96 ΕΟΚ και της απόφασης 2007 καθώς της Επιτροπής. Πού είστε εδώ πέρα, μάλιστα. Ε, κοιτάξτε, και εγώ είχα σπουδάσει γεωπόνος και πάντα μας φόβιζε η βιοχημία γιατί πηγαίναμε εκεί πέρα στην εξεταστική με, με φόβο Θεού. Και φοβόμασταν τι θα μας ρωτήσει ο καθηγητής. Οπότε ε, ευτυχώς, ευτυχώς δεν εξετάζομαι σήμερα από σας, είμαι πρόεδρος. Λοιπόν, έχετε τώρα τον λόγο. Παρακαλώ λοιπόν να μας παρουσιάσετε την ε, κατάσταση. Ευχαριστώ. Και σας ευχαριστώ και για την ευκαιρία που μας δίνετε να παρουσιάσουμε τα πράγματα. Στόχος μας είναι λοιπόν ε, να διασφαλίσουμε τους σωστούς ε, κτηνιατρικούς ε, και φτωγειονομικούς ελέγχους στα σύνορα της Ένωσης. Εδώ πέρα μιλάμε μόνο για το είδος δροσόφυλλα μελανογάστερ, όχι για άλλα είδη μήγας ή εντόμων γενικώ, αλλά μόνο για το συγκεκριμένο είδος. Η δροσόφυλλα μελανογάστερ είναι ένα είδος ε, το οποίο δεν μεταφέρει ασθένειες και δεν έχει ασθένειες ε, λόγω ακριβώς της ε, φυσιολογίας της. Η βιοιατρική έρευνα στην Ευρώπη έχει πληγεί από την απαγόρευση εισαγωγής της πάρα πολύ γιατί έχουν αναβληθεί πάρα πολλές έρευνες. Ο Δόκτωρ Οκέιν του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ του τμήματος γενετικής θα πάρει τον λόγο και θα μας παρουσιάσει ακριβώς ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Έχουμε υποβάλει πάρα πολλά παραδείγματα στην Επιτροπή σας ε, για το πόσο μας χρειάζεται αυτή η μίγα. Πρέπει επίσης να πούμε πως ε, η αντιμετώπιση διαφέρει από αεροδρόμιο σε αεροδρόμιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, παραδείγματος χάρη έχουμε και αυτά τα οποία σας έχουμε ε, αναφέρει. Ό,τι φτάνει στη Βιέννη με DHL ε, αποστέλλεται πίσω. Ό,τι όμως έρχεται με FedEx περνάει ανεξέλεγκτο. Ε, και επίσης ε, ε, οι αποστολές από διαφορά κέντρα στη ΣΥΠΑ από όπου προέρχονται οι περισσότερες τέτοιες μύγες πηγαίνουν με FedEx στο Stansted γιατί εκεί πέρα, πηγαίνει, εκεί πέρα είναι το κέντρο της FedEx αλλά εκεί πέρα δεν έχουν κέντρο υποδοχής ζών σε αντίθεση με το Heathrow. Οπότε ό,τι πάει στο Stansed αποστέλλεται πίσω. Και δεν είναι καν ενιαία η αντιμετώπιση. Σε άλλες χώρες ε, πηγαίνουν τα πακέτα πίσω, σε άλλες περνάνε. Στην ε, Πολωνία ζητάνε κτηνιατρικούς ελέγχους, στους οποίους δεν μπορεί να κάνει κανείς, γιατί όπως μπορεί να επιβεβαιώσει και ο πρόεδρος, η κτηνίατροι δεν ασχολούνται ιδιαίτερα με την δροσόφυλλα μελανογάστερα, αλλά με άλογα, γάτες ε, και τέλος πάντων άλλα ζώα. Οπότε δεν υπάρχουν ε, ειδικοί οι οποίοι μπορούν να κρίνουν την κατάσταση της υγείας της μήγας αυτής. Έχουμε και άλλα παραδείγματα αποστολών ε, πακέτων δηλαδή που γύρισαν πίσω χωρίς να ανοίξουν περίμεναν διάφορα γερμανικά πανεπιστήμια μάτια να λάβουν τα πακέτα τους. Το 2014, παραδείγματο χάρη από το Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο, είχαμε 14 αποστολές οι οποίες επιστράφηκαν χωρίς να ανοίξουν ε, λόγω κάποιας υποτιθέμενης παραβίας των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η μη ενιαία αντιμετώπιση, όσο γνωρίζω, παραβιάζει την ενιαία αγορά και την ιδέα, το σκεπτικό της ενιαίας αγοράς. Τέλος, μια προσωπική παρατήρηση. Εγώ άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά και τους ε, προηγούμενους ομιλητές και πραγματικά απορώ πως ε, με τους ε, πάρα πολύ εντατικούς ελέγχους της δροσόφυλλα μελανογάστερ μιλάμε για αποστολές που πάνε από ελεγχόμενα κέντρα και πάνε σε εργαστήρια και ασχολούνται με αυτό και από την άλλη από ό,τι φαίνεται, όπως είπαν και οι προηγούμενοι αναφέροντες, μπαίνουν εδώ πέρα διάφοροι βλαπτικοί παράγοντες και ζυζάνοι ανεξέλεγκτοι στην ε, Ένωση. Τώρα θα δώσω τον λόγο στον Δ. Οκέιν από το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ε, παρουσιάσω το ζήτημα από την πλευρά ενός ερευνητή. Η δροσόφυλλα μελανογκάστα ζει σε ολόκληρο τον κόσμο. Από το 2010 χρησιμοποιείται ε, σε διάφορα εργαστήρια χωρίς να έχει προκαλέσει οποιαδήποτε ζημιά στους ανθρώπους ε, ή στο περιβάλλον για την έρευνα γενετικών μηχανισμών. Δύο Νόμπελ, ένα από Ευρωπαίους ερευνητές Νιούσλεν Follower από το Τίμπικεν και Χόφμον από το Στρασβούργο. Ε, βασίστηκαν ε, σε μελέτες της δροσόφυλλα, μελανογκάστερ και ε, ανακαλύπτονται κάθε μέρα νέα γονίδια τα οποία δεν ξέρουμε πώς λειτουργούν και η δροσόφυλλα μελανογκάστερ είναι πάρα πολύ χρήσιμη για να ανακαλύψουμε τι, πώς ακριβώς λειτουργούν τα γονίδια. Τα τελευταία χρόνια η ανταλλαγή γενετικών αποθεμάτων στην παγκόσμια ερευνητική κοινότητα ανάμεσα στα μέλη μάλλον της παγκόσμια παγκόσμια ερευνητική κοινότητα ε, ήταν ε, ιδιαίτερα χρήσιμη. Ήμουν στο Σικάγο την περασμένη εβδομάδα στην ετήσια συνάντηση δροσόφυλλα ε, και μας μοιράσανε να καταλάβετε δροσόφυλλα, όπως βλέπετε εδώ πέρα σας δείχνω και αναφέρθηκαν στις στα νέα είδη που υπάρχουν η Επιτροπή ισχύει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Όχι, υπάρχει πρόβλημα. Πριν από δύο εβδομάδες ε, ένας μαθητής μου ζήτησε μύγες από ένα άλλο εργαστήριο και ε, μας το έστειλαν ε, με τη FedEx και στο Στάνστετ χάσαμε την αποστολή και άλλοι μαθητές, φοιτητές μου έχουν αναφέρει παρόμοια προβλήματα. Φαίνεται λογικό όταν το παρουσιάσουμε γραπτός, αλλά δεν είναι διότι αντίστοιχα είδη που δεν είναι δροσόφυλλα ε, δημιουργούν προβλήματα και ε, στη ΣΥΠΑ και στην Ιαπωνία υπάρχουν ε, εκατομμύρια αποθέματα τα οποία όμως δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ερευνητικές κοινότητες εδώ στην Ευρώπη. υπέβαλα και μία επιστολή από τον έναν καθηγητή της ΣΥΠΑ όπου συνοψίζει πολύ καλά τις δυσκολίες που υπάρχουν με τη, τη δροσόφυλλα στην Ευρώπη. Ε, δεν υπάρχουν ε, σταθμοί ελέγχου, συνοριακού ελέγχου ε, στο Στάνστετ για τη Φέντεξ, παραδείγματος χάρη. Και ε, ακόμη και αν επιτρέπεται η αποστολή για πάλι των ε, μη εγκεκριμένων ε, πακέτων, αυτό συνεπάγεται επιπρόσθετο κόστος. Επίσης θα πρέπει να διαπιστωθεί ότι ε, υπάρχει δροσόφυλλα μέσα στο πακέτο και αυτό μπορεί να γίνει μόνο από ένα εργαστήρι. Ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο επίσης ε, επιβάλλονται τέλη για τους ε, συνοριακούς ελέγχους και αντίστοιχα τέλη εμφαρμόζονται για τα άλογα. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά τάξης μεγέθους ανάμεσα στην άλογο για αυτό που σας δείχνω τώρα. Σαν ένα μικρό πακέτο χρειάζεται κάποιος 10 ευρώ ενώ ε, για να παρακάμψει τους ελέγχους ε, τελικά χρειάζεται 200 ευρώ. Είναι απαγορευτικό το κόστος ε, για τους φοιτητές. Είναι πολύ εύκολο να κάνεις ένα κλικ στο ίντερνετ, να παραγγείλεις ένα στέλεχος και τελικά να στο απορρίψουν, να, παρα... να κολλήσεις στο Στάνστετ. Ε, και δεν μιλάμε για ε, κρυφές εισαγωγές. Ακόμη ε, και όταν γίνονται νόμιμα οι εισαγωγές υπάρχουν αυστηρότατοι έλεγχοι και αυτό είναι καταστροφή για την, τους σκοπούς της έρευνας, διότι τη δυσχεραίνουν. Ε, πολλές ε, αποστολές ε, προέρχονται από μικρά ερευνητικά εργαστήρια που ουσιαστικά μας κάνουν τη χάρη, κάνουν τη χάρη στα ευρωπαϊκά εργαστήρια για να στείλουν αυτές τις αποστολές διότι οι δοκιμές που χρειάζονται για την συμμόρφωση είναι δυσανάλογα μεγάλες σε σχέση με τον κίνδυνο που υπάρχει. Επίσης στην πράξη είναι πολύ δύσκολο να τηρηθεί και η προθεσμία 24 ωρών διότι και τα εργαστήρια έχουν δικό τους χρονοδιάγραμμα. Λοιπόν, ακόμη και με ένα αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο, οι εισαγωγές ε, με μελανοκάστες στη ΣΥΠΑ αντιμετώπισαν ε, παρόμοια προβλήματα, όμως οι αρμόδιες αρχές ε, τα περασμένα χρόνια συνεργάστηκαν με τα εργαστηρία και έτσι ε, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα πολλαπλών αδειών του εργαστηρίου υποδοχής ε, χωρίς τέλη ελέγχου δείχνει ένα αποτελεσματικό σύστημα διευθέτησης αυτού του, του προβλήματος. Θα πρέπει να δεχθούμε την αποστολή στελεχών ανάμεσα σε αναγνωρισμένα εργαστήρια εφόσον δεν υπάρχουν ε, αρνητικές συνέπειες ε, για τους ανθρώπους ε, και για το περιβάλλον. Το κόστος θα πρέπει να υπακούει στην αρχή της αναλογικότητας. Θα πρέπει να βρεθούν εφικτές λύσεις για να ικανοποιηθούν και ανάγκες της ερευνητικής κοινότητας και σίγουρα θα πρέπει να αποφύγουμε τους επαχθείς διεθνείς ελέγχους ε, και τα απαγορευτικά τέλη. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Πατρίτσια Λάνχαμερ τώρα έχει το λόγο για την Κομισιόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα. I have to say I completely agree with you. The import... Συμφωνώ. Το όλο σύστημα ελέγχου των εισαγωγών πρέπει να είναι εναρμονισμένο στα κράτη-μέλη και να λειτουργικό Κατανοούμε λοιπόν το πρόβλημά σας, έχουμε κατανόηση. Από την προηγούμενη φορά που συναντηθήκαμε σε αυτή την Επιτροπή, το Δεκέμβριο του 2013 θαρώ, ήρθαμε σε επαφή με πολλά κάτι μέλη προς ενημέρωση για να διευκρινίσουμε τι μπορεί να γίνει με τα μη εναρμονισμένα αυτά ζώα. Μη εναρμονισμένα ζώα αποκαλούνται διότι δεν έχουμε καθορίσει από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεκριμένου όρου εισαγωγή Έχουμε καθορίσει τον κανόνα ότι θα πρέπει να παρουσιάζονται σε ένα μεθοριακό σύστημα μεθοριακού ελέγχου για κτηνιατρικό έλεγχο. Ε, είπαμε ότι με, δεν πρέπει να γίνουν φυσικοί έλεγχοι στο μεθοριακό σταθμό για την υγεία των ζώων ή συγκεκριμένους ελέγχους για να δουν εάν τα ζώα έχουν, ε, είναι φορείς μορισματικών ασθενειών διότι ξέρουμε ότι έρχονται από ερευνητικά εργαστήρια ε, αυτά τα ζώα. Πρέπει να διενεργούνται οι έλεγχοι για να είμαστε σίγουροι ότι σε αυτές τις αποστολές πράγματι υπάρχουν δροσόφυλλα μελανογάστα. Έχουμε περιπτώσεις όπου ζώα με πιο, πιο επικίνδυνα όπως και για τα φυτογενειακά θέματα, όπως ακούσαμε στους προηγούμενους ε, αναφέρονται εισάγονται και διατείνονται ότι δεν παρουσιάζονται τόσο μεγάλο κίνδυνο. Γι' αυτό θα πρέπει να επαληθεύουμε, να εξακριβώνουμε ότι η παρτίδα που έρχεται από ένα ερευνητικό εργαστήριο πραγματικά περιέχει τα αναγραφόμενα. Ξέρουμε ότι περιγράψατε πολλά προβλήματα σχετικά με την ταχυδρόμηση αυτών. Και εκπλήσωμαι που ακούω ότι στέλνονται με ταχυδρομείο αυτά τα ζώα, διότι θα περιμέναμε να παραδίδονται ταχύτερα μέσω των εταιριών μεταφοράς, των courier. Βλέπω ότι κουνά το κεφάλι σας. Ίσως θα έπρεπε να το συζητήσουμε αυτό διμερώς. Ε, διότι βέβαια ε, θέλουμε να έχουμε ένα πιο εναρμονισμένο σύστημα εισαγωγών και γι' αυτό θα χρειαστούμε τη βοήθειά σας όμως τούτων λεχθέντων γνωρίζουμε από τους εκπροσώπους ελέγχου εισαγωγών με τους οποίους συζητήσαμε την εισαγωγή των ζώων και με εκπροσώπους και των 28 κρατών μελών ε, δεν μας ανέφεραν τα πρόσφατα προβλήματα που παρουσιάσατε δεν μας είπαν οι εκπρόσωποι μας ότι υπάρχουν προβλήματα. Ισχυρίστηκαν τα πάντα λειτουργούν ομαλώς και τους περιγράψαμε και τους είπαμε ότι θα πρέπει να είναι γρήγοροι με τους ελέγχους όσον αφορά αυτά τα ζώα που έχουν και σύντομη ζωή, ε, κύκλο ζωής. Επιπλέον μπορούμε να σας υποσχεθούμε βέβαια ότι προβλέψαμε τη νομική βάση για παρεκκλήσεις από υποχρεωτικούς ελέγχους στα ζώντα ζώα στο σχέδιο κανονισμού για τις επίσημους ελέγχους που συζητείται στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Να σας πω όμως εξίσου ότι υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις σχετικά με τις παρεκκλήσεις διότι κάποιοι συνάδελφοι του Κοινοβουλίου δεν θεωρούν ότι δεν θα έπρεπε να διενεργούνται έλεγχοι σε οποιοδήποτε ζών ζώο. Προβλέψαμε στην νομοθεσία περί της υγείας των ζώων, κάτι που συζητείται στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο, προβλέπουμε παρέκκληση από τις απαιτήσεις περί εισαγωγής όσον αφορά αυτού του είδους τα ζώα που χρησιμοποιούνται για την έρευνα. Πρέπει να περιμένουμε την λήξη των συζητήσεων στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να περιμένουμε για την έγκριση των δύο νομοθετημάτων πριν πραγματικά να είμαστε σε θέση μέσω δευτερογενούς νομοθεσίας να προβλέψουμε οι κανόνες. Πρέπει να κατανοήσετε ότι πρέπει οι βασικές νομικές πράξεις να παρέχουν επαρκή ασφάλεια πριν στη δευτερογενή νομοθεσία να μπορέσουμε να προβλέψουμε απλουστευμένες και ε, εναρμονισμένες διαδικασίες. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. για την συζήτηση αυτή με την Κομισιόν. Και θα ήθελα να πω πως αυτό το οποίο μας είπε η Κομισιόν είναι πολύ πιο θετικά από αυτά τα οποία μας είχε πει στο παρελθόν. Δεδομένης δε της κατάστασης και του ενδιαφέροντος που έχουμε δει, κάποια στιγμή φοβάμαι πως ε, θα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτή την ε, διαδικασία. κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρξει μια σφραγίδα η οποία θα ισχύει από άκρη σε άκρη της ε, διαδικασίας από το ένα εργαστήριο στο άλλο. Για ε, να μην είναι τόσο δίσκαμπτη η διαδικασία. Ή τουλάχιστον να υπάρχει ένα κεντρικό σημείο στην Ευρώπη όταν ε, υπάρχουν επιστημονικά φορτία από άλλη ήπειρο. Ξέρω πως είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει εξαίρεση για ένα ζώο. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι μεταδοτικό, δεν μεταδίδει αρρώστιες σε φρούτα τα οποία δεν έχουν ήδη ε, κάποιο πρόβλημα και πράγματι είναι πάρα πολύ δύσκολη η ε, κατάσταση και ξέρω τη σημασία που έχει η υδροσόφυλλα ε, για την έρευνα παγκοσμίω. και το ότι σημαίνει για την έρευνα διαφόρων ασθενειών. Θα πρέπει λοιπόν η υπόθεση να γίνεται πιο γρήγορα, να απλοποιηθεί, να υπάρχει μια ενιαία αντιμετώπιση και να είναι και αναλογική έλεγχη. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να εξαρτάται από την τύχη το εάν θα φτάσει ένα φορτίο ή όχι. Και η κυρία Γκρός ανέφερε άλλο ένα παράδειγμα. Και από ό,τι φαίνεται το ένα αεροδρόμιο τα σταματάει, το άλλο τα περνάει. Δεν ξέρω, μπορεί να χαίρονται κάποιοι ερευνητές κάπου, αλλά δεν είναι η κατάσταση αυτή. Οπότε εγώ θα χαιρόμουν ε, να υπάρξει κάποια βελτίωση. Και θα πρέπει επιτέλου και η Ευρώπη να ανταποκριθεί στο ρόλο της αν είναι να γίνεται σοβαρή έρευνα εδώ πέρα ή να διατηρηθεί η δυνατότητα αυτή, αλλά... Κοιτάξτε, αν έχουν ε, τα, τα εργαστήρια ή τα πανεπιστήμια πρόβλημα σε μία χώρα και σε άλλη όχι, προφανώς είναι στρέβλωση και του επιστημονικού ανταγωνισμού, έτσι. Και βεβαίως εδώ πέρα παραβιάζεται και η αρχή τη εσωτερική αγορά. Πρέπει λοιπόν να δράσουμε γρήγορα και αυτό το οποίο θα συμβούλευα εδώ πέρα του αναφέροντε είναι να ξανασκεφτούν μήπω ε, κάποιοι από του ε, επιφανεί επιστήμονε που αναφέρατε, του ε, νομπελίστες, να μαζευτούν εδώ πέρα και να συναντηθούν με βουλευτές, με συντονιστές κοινοβουλευτικών ομάδων που από ό,τι φαίνεται δυσκολεύονται να αντιληφθούν ε, την ε, ε, επιστημονική σημασία αυτής της υπόθεσης. Έτσι για να κάνετε κάτι από την πολιτική πλευρά. Αλλά δεν θεωρώ πως εμείς πρέπει να περιορίσουμε την πίεση αυτή. Ακόμα και για ένα ζώο να, να πρόκειται για ένα συγκεκριμένο είδος, νομίζω πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτή η υπόθεση. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Θα δώσω ξανά τον λόγο στους ε, αναφέροντες και πείτε μας ε, τι γίνεται. Είναι παντού τα ίδια τα προβλήματα. Α, ο κύριος Βίλαντ. Κοιτάξτε, από ό,τι φαίνεται η κατάσταση εξαρτάται τελείως από το πού θα πέσει κανείς έτσι, και το, το τι θα του τύχει. Αυτή είναι, αυτό είναι το καθιστός. Έχει τον λόγο. Μάλιστα, να επαναλάβω στην κυρία Λάγκχαμερ. Κοιτάξτε, είναι προφανές αυτό το οποίο είπαν και οι βουλευτές. Ε, κάποια στιγμή πρέπει να ασχοληθούμε λίγο σοβαρά και με τα θέματα αυτά της έρευνας και ε, να δούμε εάν και κατά πόσον είναι επικίνδυνη η δροσόφυλλα μελανογκαστέρε. Δεν είναι έτσι, να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Και εμείς ε, ευχαρίστως να συνεργαστούμε με την Κομισιόν και να σας ε, πληροφορήσουμε για τα πάντα. Κοιτάξτε, να σας πω πως ε, όσον αφορά το αεροδρόμιο της ε, Φραγκφούρτης και τα τέλη, Είμαστε σε δικαστική διαμάχη και το Διοικητικό Δικαστήριο της περιοχής κατέληξε στο ότι ήταν πάρα πολύ χαλαρή η κτηνιατρική έλεγχη και τι κάνουνε, περνάνε τα πακέτα και τσεκάρουν ένα κουτάκι το οποίο λέει υγειονομική κατάσταση καλή. Εν τω μεταξύ τα ζώα έχουν πεθάνει, άλλα είναι πτώματα μέσα. Δηλαδή δεν να πείτε ότι και κάνουν και κανένα σοβαρό έλεγχο. Α, όπως σας είπα είμαι στη διάθεσή σας. Εγώ μπορώ να σας αναφέρω όλες τις περιπτώσεις που γνωρίζω για να βρούμε μια λύση κάποτε λογική. Ε, πρέπει να πω ότι δεν κατάλαβα ακριβώς τη λογική που της απάντησης που μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακόμη και αν υπήρχε μια εξαίρεση, ε, κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να ε, επιβεβαιωθεί το αριθμός των ε, ειδών που συμπεριλαμβάνονται σε κάθε αποστολή, σε κάθε πακέτο. Το πρόβλημα είναι ότι οι σταθμοί συνοριακού ελέγχου έχουν κατασκευαστεί, σας είπα, για άλογα και τέτοια, τέτοιου είδους ζώα. Οι κτηνιατρικές αρχές δεν θέλουν να βάλουν τέτοιο σταθμό στο Στάνσετ διότι λένε ότι θα κοστίσει εκατομμύρια λίρες γιατί εξ ορισμού ο σταθμός συνοριακού ελέγχου μπορεί να χειριστεί όλα τα ζώα. Προτείνω λοιπόν ε, με προσοχή να εξετάσετε τις ε, ρυθμιστικές ε, διαδικασίες της ΕΥΠΑ. Μπορεί να μην είναι εφαρμοστές όλες στην Ευρώπη, όμως σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα μπορεί να βρεθεί ένας τρόπος ε, του ζητήματος χωρίς ε, αυτό να συνεπάγεται μια ε, ακριβή διαδικασία. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε ένα συγκεκριμένο αριθμό ε, διάβλων και να λειτουργήσει το σύστημα με την άδεια, με το αντίτυπο της άδεια που έρχεται από το εργαστήριο να πιστοποιείται ο αριθμός των στελεχών δροσόφιλων μονοκάστερ μέσα στο πακέτο και να μην δημιουργείται πρόβλημα. Ε, και, δεν, επίσης θα πρέπει για την πανεπιστημιακή κοινότητα να ε, προβλέπεται η κανονική συνηθισμένη ταχυδρομική αποστολή, γιατί αυτό προβλέπεται από την Ταχυδρομική Ένωση. Ε, θέλετε ξανά τον λόγο κύριε Λαγκχάμερ, γιατί υπήρξε μια ερώτηση για σας. Νομίζω αν ξεκαθαρίσει θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να επανέλθω στη, στο ζήτημα της έγκρισης ε, τον Σταθμό συνοριακού ελεγχού. Δίκιο, έχετε απολύτως. Πρέπει να υπάρχει κατάλληλη έγκριση για να γίνει έλεγχο ζών των Χρειάζεται όμως και ένα ευέλικτο σύστημα ελέγχου. Ο σταθμός συνοριακού ελέγχου δεν χρειάζεται να είναι εξοπλισμένος ε, για υποειδή, για άλλο εν πάση περιπτώσει, για να ελέγξει μύγες. Ε, ε πάντως, ε, πρέπει να υπάρχει η θέληση, να υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό, κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό, κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό, είναι κάτι που πρέπει να αποφασίσει το κράτος μέλος. Και επίσης οι αποστολές με το κανονικό ταχυδρομείο θα πρέπει να ε, περνούν από το σταθμό σωριακού ελέγχου επίσης. Δεν γίνεται όμως αυτό αν δεν φέρνουν την κατάληψή μαζί, ό,τι εμπεριέχουν δηλαδή ζώντα ζώα. Και στο παρελθόν υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις. Και τότε δεν απεστάλησαν τα ε, ζώα τα ίδια αυτά στους συνοριακούς σταθμούς αντίστοιχα. Όταν μιλάτε για τους κανόνες που ισχύουν ε, στη ΣΥΠΑ θα πρέπει να κοινοποιούνται εκ των προτέρων ε, τα ζώα στους συνοριακούς ελέγχους έτσι. Πολύ ευκολότερα οι συνάδελφοι μπορούν ε, να ξέρουν από πού προέρχεται το αίτημα με την επιστολή όταν έχουν σχέση με κάποια εταιρεία όπως η DHL ή η FedEx για να ξέρουν περί πρόκειται να φτάνει η αποστολή. Μιλήσατε για το πιστοποιητικό ε, υγείας. Τα προβλήματα στην ΒΕΝΑ, παραδείγματος χάρη, θα μπορούσαν εκ των προτέρων να έχουν ρυθμιστεί αν υπήρξε αν είχε υπάρξει ο κατάλληλος προγραμματισμός για την αποστολή του πακέτου και, τη, με, και πρώτερη ειδοποίηση ε, προς τον συνοριακό σταθμό την ιατρικού ελέγχου. Όταν οι εξαγωγείς έρχονται σε άμεση επαφή με, τα, ε, με τους εν λόγω συνοριακούς σταθμούς ε, ελέγχου δεν υπάρχει κανονικά κανένα πρόβλημα. Έχουμε συζητήσει με τα κράτη-μέλη για, τον για την εναρμόνιση των ελέγχων και την επίσπευσή τους. Θα μπορούσατε και εσείς ενδεχομένως να συστήσετε ε, στους πελάτες σας ή στις πηγές σας, δεν ξέρω πώς να τους πω, καλύτερα να προγραμματίζουν τα, τις αποστολές, ώστε να βελτιώσουμε και από τις δύο πλευρές το σύστημα. Ευχαριστώ. Ε, πρέπει να προσέξουμε μην γίνει πολύ πολύ βλακό το σύστημα όμως. Γιατί ξέρετε όπου λαλούν πολύ κοκόροι αργεί να ξημερώσει. Πρέπει όμως να έχουμε μια νομική βάση. Έμαθα εδώ πέρα πως υδροσόφυλλα, μελανογάστερ είναι ένα μην αρμονισμένο ζώο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά συζητιέται αυτή τη στιγμή μια νομική βάση για εξαιρέσεις στο Κοινοβούλιο. Οπότε δεν ξέρω ποιος συνάδελφός σας στην Κομισιόν είναι αυτός τον οποίο πρέπει να πείσουμε. Οπότε, κύριε Βίλαντ, παραμένει ανοιχτή η αναφορά και δεύτερον, θα ενημερώσουμε την Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, να δούμε σε ποια φάση βρίσκεται η συζήτηση εκεί πέρα. Και βεβαίως θα γράψουμε επιστολή και θα παρακαλέσουμε την Επιτροπή Περιβάλλοντος να έρθει σε επαφή με τους ενδιαφερόμενους εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό νομίζω να εκθέσετε τις απόψεις σας ε, και στην αρμόδια επιτροπή. Γιατί... Εντάξει, επειδή είναι έντομα και ζώντα ζώα, δεν είναι ανάγκη να καταλήγουμε σε λάθος ε, συμπεράσματα. Καλό είναι λοιπόν να τα πείτε αυτά στην αρμόδια επιτροπή που θα συζητήσει τη νομική βάση και θα λάβει την απόφαση. Η δουλειά μας εμάς είναι ακριβώς να ε, ειδοποιήσουμε την αρμόδια επιτροπή πως υπάρχει ένα πρόβλημα. Το απευθύνουμε εμείς με επιστολή. Πρέπει να έρθετε και εσείς σε επαφή για να μην ε, μπερδέψουμε ακριβώς ε, το δικό σας το είδος με άλλα ε, τα οποία είναι επιβλαβή. Έτσι, γιατί είναι πραγματικά πρόβλημα αυτό για τους επιστήμονες. Εντάξει, αυτό θα κάνουμε λοιπόν. Φτάσαμε και στο τέλος της συνεδρίασης. Συγχαρητήρια στη γραμματεία. Πραγματικά φοβερά πράγματα λέξαμε πριν από την ώρα μας. Ανεπανάληπτες καταστάσεις. Πρέπει να σημειώσουμε την ημέρα. Αυτό αποδεικνύει την καλή προετοιμασία της γραμματείας. Οπότε εύχομαι καλό απόγευμα και ε, ο χρόνος ο οποίος ξαφνικά είναι ελεύθερος, ε, παρακαλώ να τον ξοδέψετε σωστά. Γεια σας, καλώς σας απόγευμα.